για να ξεκινήσετε τις δικές σας ψηφοφορίες. Να αρχίσουμε τώρα τις δικές μας ψηφοφορίες. είμαστε όλοι μας παρόντες για τις ψηφοφορίες. Να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά όλα τα μέλη της Επιτροπής, από όλο το Προεδρείο, από όλους εμάς και από τους, πέντε μας, και από τους πέντε μας. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Έχουμε 17 νομοθετικές εκθέσεις που μας περιμένουν. Όχι μία, ούτε δύο, 17 και 8 νομοθετικές γνωμοδοτήσεις. Μη νομοθετικές εκθέσεις 6 ε, ε, και μη νομοθετικές γνωμοδοτήσεις 5. Και μέχρι το τέλος της θητείας, κατά πάσα πιθανότητα, 15 νομοθετικοί φάκελ θα εμφανιστούν στο τραπέζι της Ήτρε. Έρευνα. Κόσμε, Κοπέρνικους, ε, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, ε, δορυφορικές επικοινωνίες, ενέργεια, κάποια νομοθετικά, κάποια νομοθετικά θέματα, προτάσεις, ε, διάστημα, ε, νομοθετική πρόταση για τις δορυφορικές επικοινωνίες, πάρα πολλές προτάσεις όπως βλέπετε. Επομένως, μεγάλες και πολλαπλές δραστηριότητες μας περιμένουν. Έχουμε και κάποια νέα μέλη Θα αναφέρω τώρα τα τακτικά μέλη. Με αλφαβητική σειρά. EPP Romania. Από το ΕΛΚ τη, Ρουμα... τη Ρουμανία. Σας παρακαλώ σκοθείτε. Κύριε Μπουσόη, πού είστε. Α, δεν είστε εδώ. Ο προηγουμένο ήταν στην ΑΦΕ, την ΚΟ και την ΕΜΒΗ τα προηγούμενα δυόμιση χρόνια. Ο επόμενος, με αλφαβητική σειρά, η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς. Ρεμπέκα. Παρακαλώ. Ωραία, σε ξέρουμε όλοι δηλαδή. Σήκω, να σε δούμε ακόμα μία φορά. Σε ευχαριστούμε που επανέρχεσαι ως τακτικό μέλος της Επιτροπής μας. Η Ρεμπέκα Χάρμς ξεκίνησε το 2004 τη θητεία της ως τακτικό μέλος της ΣΥΤΡΕ και τα τελευταία χρόνια ήταν συμπρόεδρος των Πράσινων. Πολύ ενεργή για θέματα Ουκρανίας. Και τώρα επανέρχεται στην Ήτρε. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Κομπάτσεφ από την Βουλγαρία, σοσιαλιστής. Μόλις έχει εκλεγεί ο κύριος αυτός από τη Βουλγαρία. Ε, απόφυτος του Πολυτεχνείου της Σόφιας και αναπληρωτής ε, στην Επιτροπή Αναφορών και στην Επιτροπή Μεταφορών. Πολλή δουλειά έχετε μπροστά σας. Έχουμε και νέα αναπληρωματικά μέλη επίσης. Την κυρία Μόσκα, Ιταλ, Ιταλίδα Σοσιαλίστρια και τον κύριο Σκλέτς από τους Πράσινους, Κροάτης, τον κύριο Σμιθ πράσινο από το Ηνωμένο Βασίλειο και τον κύριο Μποργέτσιο από το ΙΕΝΕΦ. Ιταλός βέβαια. Τέσσερα αναπληρωματικά μέλη. Αυτά εν είδη ενημέρωση τα λέω στην αρχή και τώρα πάμε στη δοκιμαστική ψηφοφορία, ως συνήθως. Βάλτε την κάρτα σας στη σχισμή και αρχίζουμε την ψηφοφορία, τη δοκιμαστική προφανώς. Okay. Ε, Is okay? One EPP, e Έχουμε έναν ε, υπεράριθμο ευρωβουλευτή από το ΕΛΚΑ. Προφανώς δεν είναι νέο μέλος, γιατί δεν είναι και παρόν εξάλλου ο κύριος αυτός, που είναι υπεράριθμος. Ξεκολουθούμε να έχουμε έναν, ένα ευρωβουλευτή υπεράριθμο από το ΕΛΚ. Τώρα είμαστε εντάξει. Τέλεια. Okay, so let us go to the... Πολύ ωραία. Περνάμε στην ε, πραγματική ψηφοφορία τώρα. Η χρήση της ζώνης συχνοτήτων 470 με 790 MHz στην Ένωση. Καταρχάς, η Πατρίτσια Τόια είναι η συγγετρία. Έγινε ένας πολύ επιτυχής ε, τριμερής διάλογος, το ξέρετε. Και τώρα ψηφίσουμε. Μία φορά θα ψηφίσουμε, ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ένας από το παραπάνω πάλι. Ποιος είναι αυτός ο παραπανίσιος. Ο κύριος Μπουσόη. Ψηφίζει παρόν δεν είναι παρόν. Τώρα είμαστε εντάξει. Κλείνει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Τέλειο αποτέλεσμα. Μπράβο κυρία συγήτρια. Συγχαρητήρια σε όλους. Πάμε τώρα στην δεύτερη τελική ψηφοφορία. Σδισλάβ Κρασνοντέψκι απόφαση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη θέσμηση μηχανισμού ανταλλαγή πληροφοριών όσο αφορά τι διακυβερνητικέ συμφωνίε. Λέγεται και ΙΓΚΑ αυτή η συμφωνία, έτσι, Intergovernmental Agreement, IGA. Λοιπόν, με ονομαστική ψηφοφορία. Όχι, όχι, διορθώνει ο Πρόεδρος με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συγγνώμη. The vote is open. I close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. 50 ψήφοι πέρ, Πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια συνάδελφε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ο καθηγητής Κρασνοντέμσκι μου ζήτησε να ζητήσω συγγνώμη δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρίσκεται σήμερα γιατί συμμετέχει στην ε, προετοιμασία της επίσκεψης της Άγγελα Μέρκελ στην Πολωνία και μου ζήτησε να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές για την εξαιρετική συνεργασία και χαίρεται όλος ιδιαίτερος που όλα πήγαν τόσο καλά. Σας αποστέλει χαιρετισμούς. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στην τελευταία μας ψηφοφορία που είναι η, ε, το σχέδιο γνωμοδότησης ε, για την αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και των άλλων μορφών διακρίσεων που φύλλονται στην υπηκότητα, τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς. Η συντάκτρια γνωμοδότησης είναι η Εύα η ευα Καϊλή και θα ήθελα να περάσουμε στη συμβιβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 106 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 110 υπέρ, κατά αποχές να την ελέγξουμε καλύτερα. Ελέγχουμε ηλεκτρονικό στην 110. Έναρξη ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές. Καλύτερα να την ελέγξουμε, δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικό στη συμβιβαστική τροπολογία 6. Πέρας της ψηφοφορίας. Θεέ μου, πώς μπερδεύτηκα. Ε, τι να σας πω, να σηκώνετε καλά τα χέρια. 26, υπέρ. Κατά. Με αποχές, εγκρίνεται. Ελκ, παρακαλώ, σηκώντε τα χεράκια. 27, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 133 υπέρ. Α, ξέχασα την 28. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 135. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ήταν σαφές νομίζω. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικό στην 141. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά... Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Σαφές το αποτέλεσμα. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες, οι 150 και 37, τις ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 151 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 156 Λοιπόν, πρέπει να ψηφίσουμε και την 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι 157 και 158 και 159 είναι ε, ταυτόσιμες όλες μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. Λοιπόν, έλεγχος των ε, τριών αυτών ε, τροπολογιών. 157, 158, 159. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνονται. 161 και 162 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβεβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Να την ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 67. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αυτή τη φορά. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικώς την 6. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82-83 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19. Λοιπόν, συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99 και 16 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές, Καλύτερα να κάνουμε έλεγχο. Ψηφίζουμε την 100 ηλεκτρονικός. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Καλύτερα να την ελέγξουμε και τη 17. Πέρα στις ψηφοφορίες για τη 17. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συγγνώμη. Τι θέλετε να ελέγξουμε. Την 103 θέλετε να την ελέγξουμε. Εντάξει, να την ελέγξουμε την 103. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα με ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σύνολο του κειμένου. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά για τη σημερινή μας ψηφοφορία. Και τώρα μπορούμε, λοιπόν, τώρα, να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Έχουμε μία μικρή καθυστέρηση.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 Dear colleagues, ladies κυρίες και κύριοι, ενημέρωση σχετικά με τι ανεξελίξει διαπραγματεύσεις περιαγωγή χονδρική. η κυρία Κούμπουλα Νάτρη είναι η συγγητριά μα. Uh, Θα προσπαθήσουμε την επόμενη εβδομάδα να ολοκληρώσουμε, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι η συγγητριά μας θα μας ενημερώσει για το τι έχουμε και προς ποια κατεύθυνση οδεύουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο της Επιτροπής. Είμαστε πολύ κατηγορηματικοί στις απόψεις μας και είναι πάρα πολύ καλή η σκιώδηση. Πραγματικά νιώθω ότι κάνουμε πολύ ομαδική δουλειά και πιστεύω ότι και στον τριμερή διάλογο θα έχουμε την ίδια συνεργασία. Χθε είχαμε και τον Μαλτέζο Υπουργό για τον Αρμόδιο για τα ψηφιακά θέματα, όπου το συζητήσαμε, το θέσαμε αυτό το θέμα και αναφέραμε τον θέλουμε να εργαστούμε για τον ανταγωνισμό, για την αγορά των τηλεπικοινών και για το συγκεκριμένο θέμα που θεωρούμε ότι είναι βάση αν θέλουμε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τους καταναλωτές. Είναι ένα λεπτό από πολιτικής πλευρά ζήτημα. Έχουμε προσχεθεί ήδη εδώ και, χρόνο, και καιρό στους Ευρωπαίους πολίτες. 15 Ιουνίου το επόμενο καλοκαίρι θα υπάρχουν πλέον τέλη περιαγωγής στους λογαριασμούς της κινητής τους τηλεφωνίας. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ήθελε λίγο πιο υψηλές τιμές, κάτι διαφορετικό σε σχέση με εμάς δηλαδή, που σημαίνει ότι ο καταναλωτής ε, παραδείγματο χάρη όταν ταξιδεύει μπορεί να χρησιμοποιηθεί λιγότερο δεδομένα. Η μηδενική τιμή για τους καταναλωτές θα μπορούσε να ισχύει για τα ε, δεδομένα Στο πλαίσιο μια πολιτικής υπεχαράχθηκε το φθινόπωρο σε σχέση με την χρήση δεδομένων. Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, οι δύο διαπραγματευτέ, πιστεύω ότι προσεγγίζουμε σιγά σιγά τι θέσει μα και πιστεύω να έχουμε ολοκληρώσει, αν όχι την επόμενη Τρίτη, πάντω έγκαιρα. Ελπίζω να λάβουμε την απόφαση. Θέλουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας νωρίς, ώστε το αργότερο στον Ολομέλεια του Απριλίου να συζητηθεί το θέμα. Σας ευχαριστώ για τη μέχρι τώρα υποστήριξη. Και θα συνεχίσω. Το θέμα που μας απασχόλησε χθε και το πιο δύσκολο θέμα είναι η τιμή για το Data Cup. Μόνιμη περιαγωγή, πώς θέλουμε να αποφύγουμε κάποιος να εκμεταλλεύεται το σύστημα, σπάζοντας, ε, παραβαίνοντας τους κανόνες αλλά δεν θέλουμε και να ακολουθήσουμε μια λάθος πορεία που θα ε, παρακολύσει την ε, δυνατότητα των ταξιδιωτών να έχουν ε, πρόσβαση στη χρήση δεδομένων. Πρόεδρος, υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια προς την εισηγήτριά μας, την οποία θέλω να ευχαριστήσω, δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Επομένως, respect, πλήρη σεβασμός πλήρη εμπιστοσύνη. Ουδέμια απορία ή ερώτηση. Ευχαριστώ. Next point. Και μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σήμερα της διάταξης της Επιτροπής Ήτρε. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά την εισηγήτρια, τη Μια Πέτρα. Πολύ καλή διαπραγματεύτρια είστε. Και τώρα έχουμε τη δημόσια ακρόαση με θέμα την αναθεώρηση του πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Πολύ σημαντικό ζήτημα όπως όλοι γνωρίζετε. Το Σεπτέμβριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σημαντικές προτάσεις για τον κανονισμό Μπέρεκ και ε, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Gigabyte 5G στο πέστο πακέτο για τη στρατηγική διασύνδεση. Ήτρε η Επιτροπή μας είναι η καθήλυνα αρμόδια. Για την επίτευξη των στόχων μας θα χρειαστούν επενδύσεις της τάξης των 500 εκατομμύρια τις επόμενες δεκαετίες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πρόκληση σε ό,τι αφορά ιδίω ε, το ύψος των επενδύσεων που θα πρέπει να γίνουν. Ο νέος κώδικας θα κάνει πιο ελκυστικές τις τηλεπικοινωνίες. Θα ε, τονώσει τον ανταγωνισμό. Και κάτι πολύ σημαντικό μεταξύ άλλων είναι ότι η Κομισιόν ελπίζει βελτιώνοντας τη χρήση του ραδιοφάσματος και και με την προσαρμογή των κανόνων, την πρόσληψη κοινωνία, να βελτιώσει γενικά τις υπηρεσίες και την διασυνδεσιμότητα. Θέλω να καλωσορίσω τα μέλη του πάνελ, πέντε τον αριθμό, κάθονται στο βήμα, για το πρώτο πάνελ και έχουμε και ένα δεύτερο. Πέντε τον αριθμό συμμετέχοντες οι ομιλητές μας, αλλά δυστυχώς σύντομο χρόνο αγόρευσης για όλους έχω προβλέψει και για το πρώτο και για το δεύτερο θα τα καταφέρετε όμως. Συνολικά έχετε πολύ χρόνο όλοι μαζί. Επίσης, ενίσχυση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και του Ευρωπαίου ρυθμιστή, της Μπέρεκ δηλαδή. Αυτό το προτείνει η Κομισιόν. Και θέλουμε να έχουμε εφαρμογή των κανόνων στην νέα αγορά και να περιορίσουμε τον κατακαιρματισμό και τις ασυνέπειες που παρατηρούνται σήμερα. Έχουμε πολύ σημαντικά θέματα και πολύ σημαντικές προτάσεις. Η ε, κύριο Τελκαστίγιο είναι η συγγήτρια από την Επιτροπή μας, ο κύριος Τοσενόφσκι, ο κύριος Ζωρίνιο και ο κύριος Μπόνι. Αυτοί είναι οι συγγητές μας. Τέσσερα νομοθετήματα έχουμε να εξετάσουμε. Μεγάλη ευθύνη Μεγάλη ευθύνη μας. Και όπως είπα έχουμε δύο συνεδρίες, δύο πάνελ, πέντε ομιλητές και μετά ερωτήσεις και απαντήσεις μετά από το κάθε πάνελ. Πέντε λεπτά ο καθένας ε, εμπειρογνώμων, για το κάθε πάνελ μιλάω, και για τους συναδέλφους μου τώρα, παρακαλώ να περιορίσετε τις παρεμβάσεις στα δύο λεπτά το πολύ. Θα δούμε Πόσο χρόνο έχουμε ε, μέχρι το τέλος. Θα έχουμε τέσσερα λεπτά για το πρώτο πάνελ για τους ομιλητές και δύο για τους ε, βουλευτές. Και έχουμε τρία πάρα πολύ σημαντικά θέματα τις επενδύσεις, το ψηφιακό χάσμα και το 5G, 5G. Στο πρώτο πάνελ το θέμα είναι δίκτυα και υπηρεσίες. Κύριε Σοριάνου, εσύ θα στο πρώτος μας ομιλητής, πρόεδρος της Μπέρεκ. Το 2017 οριστήκατε, κλήγηκατε πρόεδρος της Μπέρεκ. Από ό,τι βλέπω εδώ, Είστε μηχανικός λεπικοινωνιών, έχετε αποφτήσει από το Call Polytechnique και το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας σας ήσασταν υπεύθυνος για θέματα ανταγωνισμού και τηλεπικοινωνιών. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Έχετε παρακαλώ το λόγο. First speech in our yeah. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή Ήτρε που δίνει στην ΠΕΡΕΚ την ευκαιρία να παρουσιάσει την άποψή της για την αναθεώρηση. Και όπως αναφέρατε, με καλέσατε για να παρέμβω όχι μόνο ως πρόεδρος της ΜΠΕΡΕΚ, αλλά και ως εμπειρογνώμονας, γιατί ε, είμαι στον κλάδο για 15 χρόνια τώρα. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής. Πιστεύουμε, όχι μόνο εγώ, πιστεύουμε ότι ο τομέας των τηλεπικοινωνιών ε, και η ρύθμιση σε αυτόν τον τομέα είναι στο τέλος του κύκλου ζωής του. Ο κύκλος αυτός άνοιξε πριν από 20 χρόνια. Ε, ανοίγει μια νέα εποχή για τον ανταγωνισμό. Ανοίγει ο ανταγωνισμός. Δεν πεθαίνει ο ανταγωνισμός. Ανοίγει ο ανταγωνισμό σχεδόν σε όλε τι αγορέ στην Ευρώπη και η πολιτική εντολή που έχει το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Κομισιόν και που έχει δώσει στις ρυθμιστικές αρχές ήταν ακριβώς να ανοίξουν αυτή την αγορά στον ανταγωνισμό. Και σας διαβεβαιώ ότι αυτή η εντολή, αυτή η αποστολή εκπληρώθηκε καλά. Το θέμα είναι τώρα ποιοι είναι νέοι στόχοι. Ότι η πολιτική Ποιε είναι η νέα πολιτική, οι νέε κατευθυντήριε γραμμέ που θέλουν να δώσουν οι πολιτικοί ε, στι τηλεπικοινωνίε και στι ρυθμιστικέ αρχέ των τηλεπικοινωνιών. Από το 2015, εδώ και δύο χρόνια δηλαδή, έχουμε αυτή τη νέα αποστολή να διατηρήσουμε ένα ανοιχτό περιβάλλον στο ίντερνετ. Είναι μια νέα πολιτική εντολή που μας δώσατε. Ένα άλλο θέμα ε, είναι το θέμα της περιαγωγής. Το θέμα που παρουσιάσατε προηγουμένω. Έχετε την ε, αποστολή των καθήκων να κάνετε την ε, ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών ε, κάτι απτό για τους πολίτες μέσω του roaming, της περιαγωγή. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με την ε, συνδεσιμότητα. Η Κομισιόν μας λέει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια νέα φιλοδοξία στην Ευρώπη, ούτω ώστε κάθε πολίτης να έχει μια κάποια συνδεσιμότητα, να έχει 5G, να έχει το ίντερνετ των πραγμάτων, ε, να έχει το ίντερνετ με οπτικές σύνες, πολύ δυνατό ίντερνετ δηλαδή. Αυτή είναι η νέα πρόκληση που βάζει η Κομισιόν στο τραπέζι. Εμείς στην ΠΕΡΕΚ και οι εθνικές, καθώς και οι εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές είμαστε σε φάση εφαρμογής. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω ξεκάθαρα είναι ότι η πολιτική, το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα πρέπει να θέσουν τους στόχους. Τις τελευταίες μέρες μιλάμε για την ευελιξία που χρειάζεται. Είναι ρόλος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσει τους στόχους. Πέστε τα όλα έξω από τα δόντια. Σας παρακαλώ να είσαστε αποφασιστικοί, να θέσετε καλούς στόχους, το περιμένουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μπέρεκ είναι έτοιμη να λάβει μέρος στη συζήτηση. Και σε μια δεύτερη φάση να λάβει μέρος και στην εφαρμογή. Γιατί η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική από την εποχή που έγινε η πρόταση για την ε, ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών. Υπήρχε αυτή η ιδέα ότι έπρεπε να φτιάξουμε πανευρωπαϊκή αγορά. Όλοι είχαν τον ίδιο στόχο. Το θέμα είναι τι παίχτες θα υπάρχουν σε αυτή την αγορά. Όχι μόνο τι ρυθμιστικές αρχές θα έχουμε. Τώρα, πολύ συγκεκριμένα, εάν θέλουμε να πιάσουμε αυτό το τρένο, να μην το χάσουμε, θα πρέπει να αποφύγουμε τρεις μάστιγες. Θα μπορούσα να μπω και σε περισσότερες λεπτομέρειες μετά στη συζήτηση. Η πρώτη είναι ο κατακαιρματισμός, η διαίρεση. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο της ε, συνδεσιμότητας, όλοι οι παίχτες πρέπει να επενδύσουν. Δεν είναι μόνο θέμα αυτών που είναι ήδη στην αγορά ε, σε αντιδιαστολή με τους εναλλακτικού ας πούμε, παρόχους. Όλοι πρέπει να επενδύσουν. Θέλουμε ανταγωνισμό. Δεύτερη, η δεύτερη μάστιγα που πρέπει να αποφύγουμε είναι η αβεβαιότητα. Θα πρέπει. Πέντε λεφτά. Φτάσατε στα πέντε λεφτά, λέει ο κύριο Μπουζε, παρεμβαίνοντα. Θα πρέπει να εξασφαλίσετε αντικειμενικότητα, να εξασφαλίσετε την αντικειμε... ισοτιμία, συγγνώμη, μεταξύ όλων των επιχειρηματιών. Και η τρίτη μάστιγα είναι η γραφειοκρατία. Πρέπει να την αποφύγουμε. Θα πρέπει να λύνουμε τα προβλήματα, θα πρέπει να ε, βρίσκουμε καλές λύσεις. Και αν το βλέπουμε το πράγμα έτσι όλοι, νομίζω θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικά θα τρία. Δεν είναι εύκολο να σεβαστείτε και το χρόνο που σας έχω δώσει τα τέσσερα λεφτά. Τουλάχιστον όμως στην αρχή θα είμαστε αυστηροί. Ε, δίκτυα και υπηρεσίες είναι, το επόμενο, είναι αυτό το θέμα. Και το επόμενο πάνω θα μιλήσει για τη διακυβέρνηση. Σοβαρή διαφορά. Όλοι να μην ξεχνάμε το θέμα, όλοι οι ομιλητές. Δίκτυα και υπηρεσίες. Η κυρία Φουρ. Οι ευρωπαϊκές ε, τηλεπικοινωνίες και οι οργανώσεις των ε, ε τηλεπικοινωνιών ε, θα ακούσουμε τώρα την κυρία Φουρ που είναι ε, διευθύντρια στη Δανία σε μια τέτοια οργάνωση. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Δανέσκο Υπουργείο Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Έχει 10 χρόνια εμπειρία. Έχετε το λόγο. Κύριε Μπούζεκ, αγαπητοί ευρωβουλευτές. Η οργάνωση των τηλεπικοινωνιών ε, δημιουργήθηκε το 1992. 41 μέλη έχουμε και παρατηρητές. Είμαστε ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρονικών ε, υπηρεσιών ε, στην Ευρώπη. Οι περισσότερες από τις εταιρείες μας είναι ήδη στη δική τους αγορά, έχουν ήδη μπει, αλλά αντιμετωπίζουν προκλήσεις και σε άλλες και θέλουν, ενδιαφέρονται και για άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε για να εκφράσουμε τις απόψεις μας και χαιρόμαστε για αυτή την ευκαιρία. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο που υπέβαλε, το οποίο είναι καλή αφετηρία για να καταλάβουμε τη φιλοδοξία για το project αυτό, το Gigabit. Τώρα, για την ουσία του κώδικα, θα ήθελα να σας διαβιβάσω τρία μηνύματα. Καταρχάς, οι εταιρείε που συμμετέχουν στην οργάνωσή μας δεσμεύονται απέναντί σας σήμερα να φτιάξουν ε, παντού ε, πάρα πολύ γρήγορη συνδεσιμότητα οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Κανένας Ευρωπαίος δεν πρέπει να μείνει εκτός. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις ε, στην ευρυζωνικότητα είναι μια ιστορική πρόκληση. Είναι προϋπόθεση για να καταφέρουμε μια ε, πλήρη κάλυψη για όλους. Η ρύθμιση έχει πολύ λεπτό ρόλο να παίξει εδώ και μπορεί να τονώσει τι επενδύσει ή μπορεί να τι σκοτώσει, να τι καταπνίξει. Τρίτον, οι ευρωπαϊκέ επικοινωνίε μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερε επιλογέ ε, για του ευρωπαίους καταναλωτέ ε, ψηφιακών ε, υπηρεσιών. Αλλά οι ρυθμίσει και οι κανόνε πρέπει να επιτρέπουν αυτόν. Χρειαζόμαστε χώρο για να αναπτύξουμε την καινοτομία και στην Ευρώπη. Επίση, από τη σκοπιά των πολιτών και των δικτύων τώρα. Γιατί πρέπει να επενδύσουμε στο gigabit και γιατί έχει σημασία για του Ευρωπαίου. Η πρόσβαση σε πολύ γρήγορο ίντερνετ σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Νέες ευκαιρίες δουλειά. Ε, καλή ψηφιακή υποδομή, ούτω ώστε να φτιάχνουμε επιχειρήσεις ε, ε σε επίπεδο πληροφορικής. Ε, τι, τι επενδύσεις χρειαζόμαστε. Ε, υπάρχουν διαφορετικά νούμερα που ακούγονται. Πάντως υπάρχει μία σύγκληση. Ε, η πρόκληση είναι τεράστια. Αυτό, σε αυτό συμφωνούν όλοι. Η Κομισιόν ε, μίλησε για 500 δισεκατομμύρια για την ε, κοινωνία του Gigabit. Ενώ η συμβουλευτική ομάδα της Βοστόνης, που είναι κονσάλτα, α πούμε, μιλάει για 660 δισεκατομμύρια. Οποιοδήποτε και είναι το νούμερο, και οι δύο συμφωνούν ότι το μεγάλο κομμάτι πάνω από 90% θα πρέπει να προέρχεται από το ε, ιδιωτικό τομέα, ιδιωτικά κεφάλαια. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ευρωπαϊκός τομέας τηλεπικοινωνιών θα πείσει του επενδυτές να κάνουν αυτές τις επενδύσεις εάν οι ρυθμίσεις ε, είναι τεχνολογικά ουδέτερε και αν όλα τα ε, μοντέλα επενδύσεων προωθούνται παράλληλα. Η αρχή που διέπει τις ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες είναι ότι οι πάροχοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ευρυζωνικότητας με βάση την ε, τοπική αγορά. Ε, όλες οι τεχνολογίες, οπτική είναι μέχρι το πεζοδρόμιο ε, και μέχρι το σημείο που είναι ο χρήστης, ε, θα κάνουν τους στόχους του gigabit ε, πραγματικότητα και θα πρέπει με ουδέτερο τεχνολογικά τρόπο να προωθηθούν. Ο κώδικας αυτή τη στιγμή προωθεί μοντέλα συνεπενδύσεων. Πιστεύουμε όλες, ε, όλα τα κλασικά μοντέλα επενδύσεων από τους μεμονωμένους παρόγους θα πρέπει και αυτά να προωθηθούν, να μην αποθαρρυνθούν. Πιστεύουμε ότι η τεχνολογική ουδετερότητα και τα κίνητρα προ όλε τι ε, επενδύσει είναι πολύ σημαντικά, είναι από τον νόμο Κάνεφ, ούτω ώστε όλοι οι όλες οι επικράτες να καλύπτονται, όλοι οι Ευρωπαίοι να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κοινωνία του Gigabit. Πιστεύουμε ότι κάποιε ρυθμιστικέ προποθέσει μπορούν να εξασφαλίσουν αυτό το πράγμα. Καταρχά, είναι σημαντικό να γνωρίσουμε ε, το βασικό ρόλο του ανταγωνισμού για τις επενδύσεις. Ε, ένας υγιής και έντονος ανταγωνισμός είναι προϋπόθεση για την ε, καινοτομία και τις επενδύσεις. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τον ανταγωνισμό όμως με τις ρυθμίσεις και τους κανόνες. Δεύτερον, χρειαζόμαστε διατάξεις, ούτως ώστε να προωθούν οι επενδύσεις και να μην παγώσουν. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε να χαρτογραφήσουμε τα μέτρα τα οποία μπορούν να προωθήσουν τις τηλεπικοινωνίες, ε, να ε, βάλουν στο άρθρο 22 ε, τα νέα επενδυτικά του σχέδια ή στο άρθρο 59.3 για, για την κινητή κινητές υπηρεσίες, κινητή, κινητές τηλεπικοινωνίες. Πριν κλείσω και επειδή δεν έχω χρόνο, θα ήθελα να σας πω ότι χρειαζόμαστε τι ρυθμίσει, τους κανόνες, να δούμε τι κανόνες διέπουν τις υπηρεσίε. Υπάρχει προστασία ε, από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, δεν θα πρέπει όμω εδώ να έχουμε διπλή ε, νομοθεσία για να καταπνίξουμε την καινοτομία των υπηρεσιών. Επίσης θα πρέπει να έχουμε συνεπή προστασία των ακανοτών σε όλη την αλυσίδα αξιών. Με δύο βασικά βήματα μπορούμε να πετύχουμε διτό στόχο. Μπορούμε να, αυξήσουμε την επιλογή στον ανταγωνισμό και μπορούμε να προωθήσουμε τις ε, επενδύσεις. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο κύριος Μπούζεκ, δεν είναι εύκολο να σας σταματάω με τα τέσσερα λεπτά, αλλά θα το κάνω. Όλο και με μακρηγορούμε, σας καταλαβαίνω, έχετε τόσα πολλά να πείτε όμως. With, with our members, so I feel... Τόσα πολλά να πείτε στους ευρωβουλευτές, αλλά είμαι αναγκασμένος να σας διακόψω. θα μπορέσετε ενδεχομένω να κάνετε και επιπρόσθετα σχόλια μετά, μετά τις ερωτήσεις. Συγγνώμη σα διακόπτω πάντως. Επόμενος ομιλητής μας, Πίτερ Όλσον, αντιπρόεδρο και επικεφαλής ε, των ευρωπαϊκών υποθέσεων ε, του αγραφείου Έριξον ε, στις Βρυξέλλες και είναι επίσης πρόεδρος της Digital Europe, εκπροσωπεί τον ψηφιακό κλάδο της Ευρώπης, έχει λάβει εκπαίδευση στη Γαλλία και επίσης έχει μάστερ στο Royal Institute of Technology της Σουηδίας. Έχετε το λόγο κύριε Όλσον. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε για δίκτυα. Οπότε θα αρχίσω δείχνοντάς σας ε, μία εικόνα των δικτύων και νομίζω ότι είναι σωστό να τίθεται τα πράγματα σε σωστή προοπτική. Λοιπόν, όταν μιλάμε για ε, υπηρεσίε ηλεκτρονικέ ε, τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του 5G, μιλάμε για μια κοινή προσέγγιση και ένα πλαίσιο το οποίο αφορά την ψηφιοποίηση και την ε, μετατροπή της κοινωνίας ε, και του κλάδου. Γιατί είναι μια, και αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι μεγαλύτερη αλλαγή από αυτή που προβλέπαμε και πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ μακριά στο μέλλον ε, όταν κάνουμε τις προτάσεις. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή τη. Έχουν σε κάποιο βαθμό ε, καταλάβει ότι πρέπει να είμαστε διορατικοί, όμως δεν είναι μόνο το ζήτημα της επόμενης γενεάς, μια νέα γενεά ε, μετάβασης από το 4G στο 5G. Είναι μια κοινή πλατφόρμα που αναπτύσσεται παράλληλα και που δίνει τη δυνατότητα της μετατροπής πληροφορίας ε, ε, των υπολογιστών και συνεπώς η μελλοντική κατάσταση θα είναι διαφορετική από την τρέχουσα. Οι λειτουργικότητες, ε, η κατάσταση θα θα, είναι αρκετά διακρι, διακριτή από τα δίκτυα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά τούτων λεχθέντων ε, θα είναι πολλές ε, υπηρεσίες ανεξάρτητες ε, από την ικανότητα του δικτύου. Και είναι σημαντικό να γίνει κατανοητή αυτή η σχέση μεταξύ υπηρεσιών και δικτύων. Είναι επίσης σημαντικό να καταλάβει κανείς ότι το 5G και τα δίκτυά του θα συμπεριλάβουν διάφορες μορφές τεχνολογίες και, και σταθερές και ασύρματες και 4G LTE ε, η οικοδόμηση των αυριανών δικτύων ε, θα είναι πάρα πολύ εντατική και χρειάζονται επενδύσεις και ούτως ή άλλως αυτό το καλύψαμε ήδη. Αυτό σημαίνει ότι το εισόδημα, τα έσοδα από τους καταναλωτές δεν θα είναι επαρκή για να καλύψουμε τις επενδύσεις αυτές. Θα εξαρτηθεί και από την έγκριση των ψηφιακών τεχνολογιών ε, στην κοινωνία ε, και στον κλάδο γενικότερα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να σκεφτεί κανεί πέρα από τους καναλωτές ε, ευρύτερο, την ευρύτερη κοινότητα χρηστών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα είναι το κατάλληλο, να υποστηρίζουμε την ευρεία έγκριση και να συμπεριληφθούν όλοι οι παίκτε τη αγορά. Δύο σημεία θα ήθελα να αναφέρω από απόψεως δικτύωσης που είναι πολύ ε, σημαντικά νομίζω και θα ήθελα να ε, επανέλθω και σε μερικά ζητήματα. Το θέμα είναι η ουδετερότητα του δικτύου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό φαίνεται να είναι θεμελιώδες της ευρωπαϊκής πολιτικής όπως έχει φανεί στην αγορά ε, που είναι μία από τις καλύτερες, καλύτερες αγορές ως προς την ανάδειξη νικητών όταν πρόκειται για τεχνολογία και επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται τόσο ραγδαία, ε, είναι πολύ δύσκολο να ε, περιορίσει κανείς ε, το είδος της τεχνολογίας που θα εξελιχθεί στο μέλλον. Όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει επαρκή έμφαση στην τεχνολογική ουδετερότητα. Από την άλλη πλευρά, ένα ακόμη σημείο που αφορά τα δίκτυα είναι η διάθεση του φάσματος. Δεν θα υπάρξει 5G αν δεν υπάρχει φάσμα για το 5G. Είναι πολύ καλό το ότι ε, φτάνουμε κάπου όσον αφορά ε, τα 700 MHz, όμως χρειάζεται, ανά, χρειάζεται μεγαλύτερο φάσμα ε, για την ευρύτερη κάλυψη, αλλά και για τις πόλεις και για την χρήση σε εσωτερικούς χώρους είναι διαφορετικό τα 4, 5, 6 γίγα και διαφορετικό τα 23. Χρειάζεται λοιπόν να διατεθεί περαιτέρω φάσμα για να μπορέσει να διανεμηθεί μεταγενέστερα στους παίκτες της αγοράς. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε. Τώρα, θα ήθελα να πω και ορισμένα πράγματα για τις υπηρεσίες. Θα υπάρξουν ε, πολλές ε, διαφορετικές χρήσεις του 5G όταν σκεφτόμαστε την πτυχή των υπηρεσιών και θα καλύπτουν βεβαίως όλες τις υπηρεσίες που γνωρίζουμε σήμερα, τις παραδοσιακές και βεβαίως ε, η ραγδαία αναπτυσσόμενη υπηρεσία θα είναι το βίντεο και θα εξακολουθήσει. Επομένως ε, τα μέσα, το βίντεο θα εξακολουθήσουν να είναι πολύ σημαντικά, σημαντική τομής ε, και είναι σημαντική ικανότητα ε, τηλεφόρτωσης, ε, του downloading. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν μιλάμε για ψηφιοποίηση της τεχνολογίας θα υπάρξουν και άλλες απαιτήσει που το υπερβαίνουν αυτό. Και αυτό καθιστά πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάποιες υπηρεσίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του δικτύου, άλλες λιγότερο. Και πρέπει να καταλάβουμε και τη σχέση μεταξύ των δύο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τη φύση αυτών των διακριτών υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο τέταρτος, η τέταρτη ομιλήτριά μας, η κυρία Φελίση Αντώνιο, η οποία ε, είναι επικεφαλής πολιτικής του FastWeb, έχει εμπειρία στην ρυθμιστική πολιτική και μέσω του Fastweb στο, στην προσφορά ε, Triple Play στη χώρα της, ε, στην Ιταλία ε, που είναι μεγάλος παίκτη του κλάδου τηλεπικοινωνιών και επίση έχει εργαστεί για την Ιταλική Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, βουλευτές για την πρόσκληση. Fast Web ε, είμαστε υπερήφανοι που ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε τι είμαστε, τι κάνουμε για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες και για να σας παρουσιάσουμε επίσης την θέση και κάποιων άλλων εταιριών που έχουν παρόμοιες θέσεις, παρόμοιες απόψεις. Fast Web δεν είναι μόνο ένας από τους μεγαλύτερους ε, φορείς ε, παροχής εναλλακτικής ευρυζωνικότητας στην Ιταλία. Έχουμε ένα δίκτυο εφοπτικών ενών, 7,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ε, έχουμε προμηθεύσει με διαδίκτυο και έχουμε επενδύσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτή την προσπάθεια και συνεχίζουμε. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι στα σχέδιά μας και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερως ικανοποιημένοι με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το όπως είπε και ο κ. Σοριάνο, το θέμα δεν είναι πλέον η σημερινή και η εναλλακτική πάροχοι είναι να δούμε ποιοι επενδύουν και ποιοι δεν επενδύουν από αυτούς τους παρόχους. Και όπως καταλαβαίνετε πρέπει αυτοί που επενδύουν να πάρουν κίνητρα. Γιατί δεν το κάνουν μόνο για το όφελο των εταιριών τους, αλλά για τη δημιουργία και των καλών πρόσφορων συνθήκων που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντλήσει όφελος και να έχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα ο κλάδος. Φυσικά και υπάρχει πολλής δρόμος για το Κοινοβούλιο η πρόταση αυτή είναι καλή, αλλά χρειάζεται πλέον ε, περαιτέρω επεξεργασία. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις που ίσως να θέσουν σε κίνδυνο κάποια από τα πολύ σημαντικά ε, στοιχεία που έχουν οδηγήσει στην μέχρι τώρα άνθηση αυτού του τομέα στην Ευρώπη. Ο ανταγωνισμός ε, είναι ε, θα έλεγα το μόνο κίνητρο για επενδύσεις. εταιρείε επενδύουν επειδή νιώθουν την ανάσα ε, των άλλων εταιρεών στο σβέρκο τους. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θα ήθελα να περιοριστώ σε λίγα πρακτικά παραδείγματα. Σε ό,τι αφορά τις βελτιώσεις ε, της ήδη πολύ καλής αρχικής πρότασης της Κομισιόν και θα ξεκινήσω με την ιδέα της απλούστευσης του εφιστάμενου ρυθμιστικού πλαίσιου. Συμφωνώ. Η απλούστευση δεν πρέπει να γίνει απορρίθμιση. Θα πρέπει να, παρα, ε, την, να διατηρηθεί η, η ρύθμιση. Εμείς έχουμε μια πολύ προοδευτική προσέγγιση. Όταν υπάρχει μεγαλύτερη όρεξη, αν θέλετε, για βριζονικότητα, προχωρούμε οπτική να προς το πεζοδρόμιο. Κάνουμε τα 100 μέτρα δηλαδή από το κάμπινετ στο κέρμπ που λέμε και ε, Έχουμε επίσης προβεί και σε μια ε, άσκηση χαρτογράφησης. Θέλουμε να δούμε ποιοι είναι οι φορείς στην αγορά Για να δούμε, χρειάζεται ρύθμιση τελικά ή δεν χρειάζεται. Και τελικά το αποτέλεσμα είναι ψευδός θετικό αν θέλετε. Δηλαδή χάνεται η εικόνα και δεν ξέρουμε τελικά πού να οικοδομήσουμε τη στρατηγική μας, πού να την εδράσουμε. Ένα άλλο παράδειγμα είναι επενδύσεις να μην συγχέονται με εμπορικέ συμφωνίες. Συμφωνούμε ότι οι επενδύσει από κοινού μπορεί να οδηγήσουν σε απλούστευση και απορρίθμιση. Γιατί οδηγεί μια κατάσταση που έχουμε δύο φορεί και παραπάνω που έχουν ο καθένα το δικό του δίκτυο. Άρα τι θα πει αυτό, δημιουργούμε ένα σταθερό έδαφο για έναν ανταγωνισμό βάσει των υποδομών. Δεν νομίζω ότι η εμπορική συμφωνία έχει το ίδιο Γιατί ουσιαστικά δημιουργείται ένα operator, ένα φορέα που επενδύει και ο άλλο είναι εξαρτώμενο από το δεύτερο, από τον πρώτο μάλλον. Επομένω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Thank you very much, madam. Ευχαριστούμε. Ο επόμενο ομιλητή του πρώτου πάνελ, ο πέμπτο, ο κ. Φόξ Ρόμλι, αναλυτή του Global Telecoms. Και αναλυτής του City. Έκανε διάφορες ε, σχετικές αναλύσεις το 2005 και 2006. Ε, έχει ένα μάστερ στη φυσική από το Imperial College στο Λονδίνο. Ε, ε, είναι αναλυτή ε, αναλύει τις, τα αποτελέσματα διαφόρων επενδύσεων. Δεν κάνει ο ίδιος επενδύσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε για να σας μιλήσω για το νέο κώδικα ε, για τις τηλεπικοινωνίες. Ε, οι κανόνες είναι τεράστια σημασία θέμα για τι τηλεπικοινωνίε, για να έχουμε καλύτερε υπηρεσίε, καλύτερη κάλυψη κτλ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ουσιαστικέ επενδύσει σε δίκτυα ε, σε πολυετή βάση, είναι ε, για πολλές δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ε, κανονιστικό περιβάλλον, ε, ούτω ώστε να οδηγεί αυτό φυσικά σε επενδύσει. Εγώ, ω αναλυτή, μιλάω με του επενδυτέ σε καθημερινή βάση για αυτά τα θέματα και αυτό που θα προσπαθήσω είναι να σα ε, διαμηνήσω πώ βλέπουν τον κλάδο ε, και πώ ε, μπορούν ε, να προωθηθούν οι περαιτέρω επενδύσει. Κατά τη γνώμη μου. Οι επενδυτέ καταρχά θα πρέπει να έχουν καλά κέρδη, γιατί αλλιώ το κεφάλαιο θα πάει αλλού, σε, άλλα, σε άλλου τομεί, σε άλλε υπήρου οι επενδυτές ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουν κέρδη για τους ε, πελάτες τους. Έχουν το, την ηθική αυτή υποχρέωση. Ε, σήμερα βλέπουμε ότι ο νέος κώδικας μιλάει για ενθάρρυνση των επενδύσεων, χαίρομαι γι' αυτό, και για εξασφάλιση προβλέψιμου περιβάλλοντος. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τρία πράγματα σημαντικά. Καταρχάς, τη μεθοδολογία χωρίς διακρίσεις, που είναι θαυμάσια, που είναι ακρογωνιαίος λήθος για να βελτιώσει την αίσθηση των ε, επενδυτών ε, στον χρόνο. Δεύτερο, συνεπενδύσεις, ανάλυση της αγοράς, που μπορούν να δώσουν ευκαιρίες για να μειώσουμε το κανονιστικό άχθος. Τρίτον, ε, ο κανονισμός για τις οπτικές σύνες, που έχει θετική υποδοχή από, την, από τους επενδυτές, έχει αλλάξει πάρα, πολλές, πάρα πολλά μυαλά των, ε, των επενδυτών να επενδύσουν ε, στις σταθερές ε, τηλεπικοινωνίες. Ε, αυτό είναι πολύ πιο, θα εξασφαλίσει συνεπή εφαρμογή σε όλες τις ευρωπαϊκές αγωγές. Ε, οι επενδυτέ θα παρακολουθούν αυτές τις νέε προτάσει πολύ προσεκτικά όταν συζητήσουμε, ας πούμε, τα δίκτυα υψηλών επιδόσεων ε, η τάση να, έχουμε, ε, να είμαστε επιτακτικοί, παραδείγματο χάρη ε, να προτείνουμε συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις, παραδείγματο χάρη οπτική να μέχρι το, το σπίτι του χρήστη κτλ. είναι πολύ σημαντική. Ε, εγώ, είναι πάρα πολύ επίκαιρα επίκαιρα αυτά τα μέτρα, ούτω ώστε να φέρουν την ευρυζωνικότητα σε πολλούς ε, χρήστες ε, σύντομα, χωρίς να αποκλείονται ε, μελλοντικέ αναβαθμίσεις. Το κόστος αυτής της τεχνολογίας θα, θα απαιτήσει μεγάλες επενδύσεις, θα έχουμε διαφορετικές καταστάσεις σε διαφορετικές περιοχές και η αγορά θα αποφασίσει τι είναι καλύτερη και πιο αποτελεσματική λύση. Θέλω να περάσω στο δεύτερο θέμα, παράλληλων επενδύσεων. Θεωρητικά αυτό έχει θετικό δυναμικό, αλλά ανησυχούν οι επενδυτέ γιατί ε, θα, υπάρξουν, θα υπάρξουν πολλέ προποθέσει για τι ε, από κοινού επενδύσει. Αν υπάρχουν πολλέ προποθέσει, τότε οι νέοι κανόνε δεν θα χρησιμοποιηθούν απλούστατα και θα είναι μια χαμένη ευκαιρία. Ιδίω, καθώ έτσι όπω έχουν οι κανόνε, υπάρχει ένα κανόνα. Ε, ο επενδυτή ε, να δεσμευτεί ε, για ένα περιορισμένο αριθμό γραμμών και μετά να αποφασίσει αν θα αυξήσει τι γραμμέ. Ε, όμως, ε, αν κάποιος αποφασίσει αργότερα ε, να, να κάνει τις επιλογές του, δεν παίρνει το ίδιο ρίσκο και επομένως θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία στις τιμές που χρεώνονται για να α, λάβουμε υπόψη μας αυτή την πραγματικότητα. Επίσης, θα πρέπει ε, να υπάρχει να δούνε και λαβήν. Μια ουσιαστική μείωση δηλαδή στους κάνους και στις ρυθμίσεις. Τρίτο θέμα. ανάλυση ε, της αγοράς. Ε, πιστεύουμε ότι αν οι επενδυτές ε, υποστηρίζουν αυτή την ε, στάση των τηλεπικοινωνιών ε, και αν είναι ανταγωνιστική η αγορά λιανικής, δεν υπάρχει να έχουμε ε, πολλούς κανόνες για τη χοντρική. Ε, Παραδείγματο χάρη, γίνεται μια πολύ σημαντική καινοτομία όταν υπάρχουν συμφωνίες μακροπρόθεσμες χοντρικής. Ε, επίσης, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές και χώρες όπου ε, δεν, έχουν κυρίαρχη θέση οι, οι πάροχοι που υπάρχουν, ε, που υπάρχουν ήδη. Ε, συχνά ε, το επίπεδο είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο. πιστεύουμε ότι αν α, παρατείνουμε την διάρκεια της, των αναλύσεων της αγοράς πέρα από τα τρία χρόνια είναι πολύ λογικό. θα έχουμε προβλεψιμότητα ε, και επίσης ε, θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τα, τους χρονικούς ορίζοντες ε, με τις περιόδους αποπληρωμής των επενδύσεων που κάνει ο κλάδος, που είναι μία δεκαετία ή παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφου, στην εισηγητριά μας καταρχάς για τον κώδικο, για τις τηλεπικοινωνίες στην κυρία Καστίγιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλα τα μέλη του πάνελ. Νομίζω ότι Υπάρχει μεγάλη σύγκληση απόψεων στις αναλύσεις που μόλις ακούσαμε. Και εμείς έχουμε συζητήσει το θέμα από διάφορες οπτικές γωνίες. και στην Επιτροπή Ήτρε και στο Κοινοβούλιο και σε άλλα βήματα συζήτηση. Θέλω να πολύ συγκεκριμένη, γιατί είναι σαφέ ότι έχουμε σημαντικές προκλήσεις τι διακυβεύεται. Το είδαμε και από τις ομιλίες σας. Δεν θέλω να επιμείνω και δεν θέλω να αναφέρω όλα όσα είπατε κι εσείς. Πρέπει όμως να δούμε, αυτό πρέπει και ο Πίτερ, είναι το νέο σενάριο. σε σχέση δηλαδή και με τις εταιρείες over the top, τις επιφύσεις, υπηρεσίες που παρέχονται. Δεν ξεκίνησε τώρα η ιστορία. Απλά έχουμε νέες οδούς, νέες ευκαιρίες, νέους ορίζοντες. Θα εστιάσω σε έναν από τους τομέε που έχουμε διαφορετικές απόψεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και που η τελική προσέγγιση θα μπορούσε να επηρεάσει διαφορετικά τα πράγματα. Τι εννοώ ακριβώς. Τον νέο ορισμό των τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως προβλέπεται στην πρόταση της Κομισιόν. Φανταζομαι, γνωρίζετε όλοι, ότι κάθε εμπλεκόμενος έχει διαφορετική άποψη. Λειτουργικός ορισμός είπατε πρέπει να είναι. Και η δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται. Άλλοι όμως έχουν άλλη άποψη. Λένε ότι είναι τεχνητή διάκριση. κάποιων υπηρεσιών. Πρέπει λοιπόν Ο καθένας από εσά, αν θέλετε να μας δώσετε τις απόψει Sorry, Γιατί για μένα είναι σημαντικό το θέμα. Αλλά νομίζω και για όλους. Αν μπορείτε να απαντήσετε, θα το εκτιμήσω ιδιαίτερος. Όπως βλέπετε, είναι δύσκολο να τηρήσουμε το χρόνο για όλους, ε, όπως βλέπετε. Θα ήθελα να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση ε, των αγορών τηλεπικοινωνιών, ε, λέει ο κύριος Τοσενόφσκι. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι είπατε ότι τώρα εισερχόμαστε σε μία νέα γενεά και ότι πρέπει να είμαστε Επιφυλακτική. Υπάρχει αυτή η ανάγκη. Εγώ θα σχολιάσω αυτά που είπε και ο εκπρόσωπος ε, του Μπέρεκ θα ήθελα να αναφερθώ όμως και στο θέμα των επενδύσεων ε, που πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλους από τη μία και από την άλλη να μην ε, επιβαρύνουμε την αγορά με πάρα πολύ νομοθεσία. Επειδή όλοι συνομιλούμε με εκπροσώπους παρόχων υπηρεσιών, Εμένα ήρθαν σε επαφή μαζί μου κάποιοι πάροχοι υπηρεσιών και είπαν ε, ότι το άρθρο 17 αναφέρει ότι ε, θα έπρεπε να υπάρχει ε, μία ε, ισότιμη διανομή μεταξύ των ε, ε, προμηθευτών και των παρόχων. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας άποψη και μετά θα, ρωτήσω, θα κάνω και κάποιες ερωτήσεις για τον οργανισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζωρίνιο. Ευχαριστώ. Για το Wi-Fi for you. Θα μιλήσω τη μητρική μου. Ευχαριστώ το πάνελ για τις εξηγήσει που μας έδωσε. Η πρωτοβουλία Wi-Fi for Europe είναι πάρα πολύ σημαντική, ούτω ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να, μπορούν, να μπορούν να θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ε, βελτιώνει με αυτό τρόπο τη ζωή τους. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα project για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ένα σημείο αναφορά, το οποίο καθιστά δυνατό οι πολίτες να χρησιμοποιούν τα gigabit και η Ευρώπη θα πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο και θα πρέπει να έχει πρόσβαση, πρόσβαση ο καθένας. Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί γρήγορα και αξιόπιστα, ούτως ώστε οι πολίτες να έχουν πραγματική πρόσβαση ε, στην ψηφιακή αγορά. Εγώ ήρθα σε επαφή με μέλη της ε, Επιτροπής των Περιφερειών, την, ε, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με πολίτες. Κοίταξε εκθέσεις που υιοθετήθηκαν ομόφωνα, όπου οι πολίτες φαίνεται ότι είναι πραγματικά ε, πολύ ανοιχτοί σε αυτή την πιλωτική εμπειρία. Θα ήθελα να ρωτήσω τους ομιλητές μας να μας πούν τι μπορούν να κάνουν, τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν, ούτω ώστε να είναι ένα σημείο αναφορά αυτή η πρωτοβουλία. Να είναι αξιόπιστη, να είναι ξεκάθαρη και να τελεσφορήσει. Αυτή και το πακέτο που συζητάμε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ο κύριος Μπόνι, υπεύθυνο για το Gigabit Society, για την κοινωνία του Gigabit και το 5G. Ευχαριστώ πολύ και για τις ε, παρουσιάσεις. Μας ενέπνευσαν δύο πράγματα. Πρώτον, καταλάβαμε ότι υπάρχουν κάποια κρίσιμα σημεία σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, γιατί η στόχη είναι σαφής. Και ένας από τους στόχους, ή μάλλον ένα από τα κρίσιμα σημεία, αφορά τον τρόπο αποφυγής κατεκρεματισμένων λύσεων και αποφάσεων. Τι θα πει αυτό. Τότε τα κρατη θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά ταυτόχρονα. Αυτό είναι σημαντικό. Τι πιστεύετε, πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτό το έργο. Δεύτερο. Ζήτηση για νέες υπηρεσίες. Ο κύριος Όλσον μας παρουσίασε ένα πακέτο νέων υπηρεσιών σε σχέση με το e-health, το 5G, νέους τρόπους μάθησης κτλ. κτλ. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα κατάλογο πλεονεκτημάτων, ωφελιών και πώς με συνεργασία των τοπικών αρχών και των κρατών μελών. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Επόμενος, επομενή στον κατάλογό μου. Η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ τη μητρική μου γλώσσα στα γερμανικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους τους εμπρογνώμονες, όλους τους ομιλητές για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Δεν θα κάνω σχόλια, αλλά και ερωτήσεις πολλές έχω, σε δύο θα περιοριστώ. Πώς θα πετύχουμε εδώ να δώσουμε ένα σύστημα κινήτρων για επενδύσεις και για το 5G πώς θα επενδύσουμε περισσότερο. Σε ό,τι αφορά αυτά τα μοντέλα συνεπενδύσεων, αυτό προτείνει η Κομισιόν αρκεί, πρέπει να το διευκρινίσουμε περισσότερο και ανέπρος με κατεύθυνση και όλα αυτά ήταν το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα, mapping, χαρτογράφηση. Διαβάζω τις προτάσεις, ε, μου ακούγεται κάπως ε, γραφειοκρατικό και βαρύ όλο αυτό. Και νομίζω ότι έχει γίνει ε, κάποιο είδος χαρτογράφηση για το που χρειάζεται ακόμα ρύθμιση ή που δεν χρειάζεται. Άρα το χρειαζόμαστε αυτό το mapping, αυτή τη χαρτογράφηση. Είναι πρόταση της Κομισιόν, αλλά έχει νόημα ή δεν έχει. Ευχαριστώ. Ε, thank you very ε, Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα στι στις ερωτήσεις σε ό,τι αφορά ε, την ε, τόνωση των επενδύσεων. Ε, χρειάζονται επιχειρηματικά μοντέλα για το 5G. Ποια είναι η αποψή σας. Έχουμε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές που έχουν μεγάλη κάλυψη με σχετικά χαμηλό κόστος. Πώς μπορούμε να το κάνουμε για το 5G και σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές 5G. Νομίζω ότι χρειάζεται ίσως όχι ακόμα, ίσως και καθόλου να γίνει αυτό το άλμα τελικά. Και επειδή είμαστε λίγο πίσω σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, ε, γιατί είναι κάπως, ε, ε, δεν είναι τόσο ασφαλής, αν συμφωνείτε. Και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά το ψηφιακό κλάσμα, χάσμα, συγγνώμη, πώς μπορούμε να το μειώσουμε, ιδίως βέβαια στην Ήπετρο, γιατί στις πόλεις όσο είναι πιο εύκολο. Άκουσα επίσης για την βιομηχανία που θα ήθελε να πάρει ένα αμερικανικό πρώτο, τόσο πάντων συζητείτε αυτό. Υπάρχει κίνδυνο και πόσο μεγάλο είναι αυτό να έχουμε παράλληλα πρότυπα. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι ένα θέμα που επίσης συζητήθηκε, η κίνδυνη για την υγεία. Και στη Γερμανία υπάρχει μεγάλη ε, μεγάλο πρόβλημα με την εγκατάσταση νέων στήλων ε, με κεραίες και καλώδια. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Ποια είναι δικά σας άποψη. Questions, quite a lot of Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Χόκμαρκ. Ε, ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις παρουσιάσεις σας. Ε, μία σκέψη πριν τις ερωτήσεις ε, σε πέντε χρόνια, με, συγγνώμη, με το 5G θα αλλάξει ο χαρακτήρας των ε, τηλεπικοινωνιών. Ε, δεν θα μιλάμε μόνο για τηλέφωνα. Θα υπάρχει μια ροή δεδομένων σε μια κλίμακα που δεν έχουμε ξαναδεί θα είναι τμήμα της ενεργού δράσης σε κάθε τομέα της κοινωνίας. Κάποτε ο ηλεκτρισμός έκανε αυτό το ταξίδι. Εγώ αναρωτιέμαι πώς θα αλλάξει τη λογική των επιχειρήσεων ε, αυτή η κατάσταση, ε, η σύγκληση μεταξύ των διαφορών υπηρεσιών, ε, οι συμφωνίες, το βλέπουμε για παράδειγμα ήδη από την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών. Πώς βλέπετε τα πράγματα από αυτήν την οπτική γωνία. ώστε να επιτύχουμε κοινέ υπηρεσίες, καλύτερη πρόσβαση, εικονικές ε, ε, υπηρεσίες, σε σύγκληση όχι μόνο μεταξύ ε, παικτών, αλλά και μεταξύ και διασυνοριακά, επειδή μειώνουμε το κόστος της περιαγωγής δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ε, καθόλου σύνορα ε, στις ε, τηλεπικοινωνίες. Πώς βλέπετε την ιδέα πανευρωπαϊκών, διασυνοριακών, τηλεπικοινωνιακών φορέων. Είναι διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Αυτό σημαίνει νέες λύσεις επίπεδο επιχειρήσεων και σημαίνει ενδεχομένως και νέα νομοθετική δομή. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις ακόμη έχω στον καταλογό μου η κυρία Κουμπούλα Νάτρη. Επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι σκιώδης η συγγήτρια για τον κώδικα για την Έριξον θα ήθελα, την Έριξον θα ήθελα να ρωτήσω, μια και είστε ένας από τους μεγαλύτερους φορείς που αναπτύσσουν τα συστήματα 5G, ε, έχουμε το, τα καλωδιακά, ε, έχουμε ε, ήδη κάποια, κάποιες υπηρεσίες, κάποια τεχνολογία στη διάθεσή μας. Εσείς είστε υπέρ τεχνολογικής ουδετερότητας. Δεν θέλουμε πάντως κανένας να είναι δέσμιος της σημερινής τεχνολογίας. Θα ήθελα λοιπόν να μου κάνετε περισσότερο τεχνικές παρατηρήσεις σε σχέση με αυτό. Για τον Μπέρεκ, τον Μπέρεκ θα ήθελα να ρωτήσω τη μεγαλύτερη διάρκεια για τη χρήση του φάσματος, επειδή δεν προτείνεται κάτι γι' αυτό. Είναι καλύτερο ο σχεδιασμός να γίνεται σε εθνικό επίπεδο ή καλύτερο είναι να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα 10 ετών. Και αν είναι 10 έτη, για παράδειγμα να δώσουμε το κίνητρο να χτίσει κανείς το σπίτι του καλύτερα και πιο μακροπρόθεσμα, μήπως αυτό τελικά είναι αντικίνητρο και κάποιος δεν το χτίσει καθόλου αν κάποιος αγοράζει το φάσμα για να αποκλείσει κάποιους ανταγωνιστές, τότε κανένας εκεί δεν παρέχει υπηρεσίες. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού. Και για τους ε, επενδυτές, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Παρουσιάζει κάποια, παρουσιάζεται κάποια, κάποια σημεία, θε, κάνετε χρηματοδότηση και των νεοεισερχομένων, γιατί οι μεγαλύτεροι καινοτόμοι δεν προέρχονται υποχρεωτικά εντός του τομέα, ε, αλλά και εκτός. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους πιο κατεστημένους φορείς εκμετάλλευσης. Ε, υπάρχει ένας κίνδυνος ότι τα παλιά χρήματα χρηματοδοτούν τους παλιούς και τα καινούργια τους καινούριου σε μερικές περιπτώσεις είναι ενεργειακές εταιρείες, ε, σε άλλες χώρες είναι ε, μικρότερες ιδιωτικές εταιρείες και κάτι άλλο σε σχέση με τους κατεστημένους ή μη κατεστημένους φορείς, το θέμα των SMPs που υπάρχουν, αλλά μερικές φορές ε, ε, απομακρύνονται άνεση, είναι ένας πολίτης και υπάρχουν πολλοί παίκτες, ε, ε, ένα δισεκατομμύριο από τη μία και δέκα δισεκατομμύρια από την άλλη. Εσείς τι προτείνετε δηλαδή, πιστεύετε ότι πρέπει να το καταργήσουμε αυτό, τι προτιμάτε δηλαδή, προτιμάτε να γίνει ένα μονοπόλιο εκ νέου. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ράιμον δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας θέσω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα για το Wi-Fi for Europe. Είμαι εισηγήτρια για αυτό το θέμα. Σκιώδης εισηγήτρια. Η Κομισιόν στο πρόγραμμά της λέει ότι το δωρεάν Wi-Fi που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ε, πολύ ταχύ. Ξέρετε όμως ότι στις περιοχές της Υπέθρου δεν υπάρχει αυτό το γρήγορο ίντερνετ. Ε, θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για το θέμα αυτό. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν θα είναι μόνο ε, μια βιτρίνα για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πόλεις που ήδη έχουν καλή συνδεσιμότητα, αλλά το πρόγραμμα αυτό να δώσει λύσεις συγκεκριμένες στα προβλήματα που έχουν οι περιοχές της Υπέθρου με τη συνδεσιμότητα. Επίσης, τι γνώμη έχετε Πιστεύετε, ότι μπορεί να υπάρχει μια γεωγραφική κατανομή ισορροπημένη. Και επίσης, αυτός ο πειραματισμός που θα είναι πολύ περιορισμένος τελικά, γιατί μιλάμε για 6.000 με 8.000 ε, δήμους και κοινότητες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ περιορισμένοι. Πιστεύετε ότι αυτό το πείραμα τελικά θα είναι ο προπομπός της ανάπτυξης άλλων υπηρεσιών και άλλων χρήσεων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μελλοντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ καλή συζήτηση, αγαπητοί συνάδελφοι. Τώρα στρέφομαι στους ε, ομιλητές. Τους παρακαλώ να απαντήσουν σε ερωτήσεις, αλλά σύντομα. Δεν ξέρω, ίσως να επιλέξει ο καθένας μια-δυο ερωτήσεις. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να συνεργαστείτε κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν ξέρω. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Όλσεν. Να πάμε στην άλλη πλευρά μετά απέναντι. Και σε μια ώρα οι απαντήσεις από την άλλη πλευρά. Σε μια ώρα. Να το κάνουμε έτσι. Ε, ε, Ο κύριος Όλσον. Φυσικά πολλές και πολύ καλές ήταν οι ερωτήσεις. Θα πρέπει να επιλέξω σε ό,τι αφορά τον ορισμό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Θεωρούμε ότι είναι προβληματικό να χρησιμοποιούνται οι προτινόμενοι ορισμοί για το conveyance ή το number-based κτλ. Αναπτύσσονται και οι υπηρεσίες ε, τάχιστα. Μπορεί κάποια πράγματα να ήταν number-based ή να είχαμε conveyance of signals, αλλά αυτά στο μέλλον ή και ήδη από τώρα παράγονται ή παρέχονται με διαφορετικό τρόπο. Και νομίζω ότι είναι προβληματικό να είμαστε άκαμπτοι στους ορισμούς, πρέπει να γίνει περαιτέρω ανάλυση. Να κάνω ένα ακόμη σχόλιο για το 5G, 5G, αυτοκινητοβιομηχανία. Υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις, πολλές διαφορετικές προτάσεις. Και πρέπει να υπογραμμίσουμε την ουδετερότητα της τεχνολογίας. Η Κομισιόν δεν θα πρέπει να επιλέξει το με ή το δε. Αυτό θα πρέπει να γίνει από τους οργανισμούς τυποποίησης. Και η αυτοκινητοβιομηχανία και η τηλεπικοινωνιακή ε, και η πληροφορική, όλοι αυτοί οι φορείς να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν μετά, γιατί αυτοί θα πρέπει να κάνουν τις επενδύσεις ε, και να δημιουργήσουν τα δίκτυα και αυτοί θα πρέπει να καθορίσουν και τα βέλτιστα δυνατά πρότυπα. Ευχαριστώ. Κύριε Σοριάνου. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά το κίνδυνο να είναι δυσκίνητος ο ε, κανονισμός, η ρύθμιση τέλος πάντων και η συνεπένδυση, πώς μπορούμε να το ορίσουμε καλύτερα. Πρέπει να αποφύγουμε εδώ μια παρανόηση. Αυτό το οποίο αποτρέπει ε, τις αποθαρρύνεις επενδύσεις σε καμία περίπτωση δεν είναι η ε, απορρίθμιση αλλά η ρύθμιση. Πρέπει να υπάρχει σωστή ρύθμιση και ξέρω ότι υπάρχει ο πολιτικός στόχος της συνδεσιμότητας. και θα πρέπει να βρούμε σε εθνικό επίπεδο με την εργαλειοθήκη που έχουμε τι θα γίνει με τους εναλλακτικού και τους κατεστημένους ε, φόρεις εκμετάλλευσης, ποιες είναι οι προ... Ε, τιμητές επενδύσεις και ποιο σχήμα θα πρέπει να ακολουθηθεί. Καλή και απορτήση, αλλά η πρόταση της Κομισιόν είναι λίγος ρλομανδίας. Ε, είναι λίγο περιοριστική δηλαδή και επειδή δεν υπάρχει απαρκής αυτονομία για την υλοποίησή της, ενδεχομένως να προκύψει ασφάλεια, ανασφάλεια, συγγνώμη, και αβεβαιότητα στους επενδυτές οι οποίοι θέλουν να, να προχωρήσουν σε πολύ ε, μεγάλη ισχύω δίκτυα. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο σε κάθε χώρα. Άρα χρειάζεται και επαρκής αυτονομία για τα 25 χρόνια. Για την έγκριση δηλαδή και για το πώς μπορούμε για το 5G οι αποφάσεις να μην λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο εφόσον δεν θα είναι συνεκτικές μεταξύ τους. Πρέπει να σας πω ότι η Μπέρεκ μέχρι σήμερα επεξεργάζεται τα ζητήματα του φάσματος και εκδώσαμε την πρώτη μας γνωμοδότηση για το σχέδιο πρότασης ε, ε, της αναθεώρησης δεν ασχολείται βέβαια άμεσα με το φάσμα. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Έχουμε συγκροτήσει και μια νέα ομάδα εργασία για την κινητή τηλεφωνία και την περιαγωγή που επεξεργάζεται ακριβώ τι λεπτομέρειε και βλέπει τι ε, καλό και τι κακό περιλαμβάνει η πρόταση τη Κομισιόν. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε την ανάγκη για τον κλάδο να έχει την ε, επαρκή ορατότητα και να υπάρχει διαφάνεια. Αλλά προς το παρόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρυστάλλινη σφαίρα για να δούμε τι μπορεί να γίνει μετά από 25 χρόνια. Ίσως χρειαστεί κάτι σαν μια διαδικασία αναθεώρησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Διευθυντρία, ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις. Πολλές ερωτήσεις είναι ενδιαφέρουσες. Όλες είναι ενδιαφέρουσες. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από αυτές. Καταρχάς, πώς θα εξασφαλίσουμε τις επενδύσεις Δύο είναι οι βασικοί στόχοι για μας. Η τεχνολογική ουδετερότητα και η υποστήριξη όλων των ε, επενδυτικών μοντέλων. Και προβλεψιμότητα στον κώδικα, τόσο ώστε να ξέρουν πού πάμε οι επενδυτές. Ό,τι αφορά την τεχνολογική ουδετερότητα, ε, έγινε μια ερώτηση για το πώς θα εξασφαλίσουμε ε, την κάλυψη των περισσότερων Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί αν έχουμε τεχνολογική ουδετερότητα, ο πάροχος ε, αποφασίζει την τεχνολογία και πώς θα αναπτύξει γρήγορο ίντερνετ. Με αυτόν τον τρόπο θα εξαφαλίσουμε πιο γρήγορη ανάπτυξη γρήγορου ίντερνετ. Για τον νέο ορισμό που ανέφερε η Πιλάρντε Καστίγιο, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ε, για την ε, σύγκληση των ε, μηνυμάτων θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα μεταξύ των μηχανών machine to machine και επίσης θα υπάρχει δυσανάλογη, ε, δυσανάλογες ρυθμίσεις και κανόνες για, τους, για τις ρυθμιστικές αρχές, μιλάω αυτό. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε το ίντερνετ των πραγμάτων, θα πρέπει οι πάροχοι να, είναι, να εμπλακούν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Και τώρα, η επόμενη μιλήτρια, η κυρία Φελίτσο ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα απαντήσω σε καμιά δύο ερωτήσει. Ε, με επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Σοριάνο. Συμφωνώ και εγώ ότι μέχρι στιγμής οι κανόνες όχι μόνο δεν έχει εμποδίσει τις επενδύσεις, αλλά ήταν και ένα πλά στην Ευρώπη. Ε, είμαστε σε καλό σημείο για να πετύχουμε τους στόχους του 2020 στην Ευρώπη, ενώπιση του 2020. Και όχι μόνο αυτό. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι που στην Ευρώπη καταφέραμε να το πετύχουμε αυτό παράλληλα με την εξασφάλιση χαμηλών τιμών. Αυτό μας το εξασφάλισε ο ανταγωνισμός. Αν δούμε τι γίνεται σε άλλες επίρους, έτσι, οι Ηνωμένες Δεν είναι ίδιες συνθήκες εκεί. Ο χαμηλός βαθμός ανταγωνισμού στην Αμερική οδήγησε σε πολύ ψηλές τιμές. Έκανε την ευρεία ζώνη υψηλής ταχύτητας ε, να κυμαίνεται σε τιμές απίστευτες σε πολλές πόλεις. Χωρίς να εξασφαλίσει σημαντικά ωφέλη στην ανάπτυξη. Επίσης, οι κανόνες και ρυθμίσεις μπορεί να φαίνονται περίπλοκοι, αλλά συχνά μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τα σημεία συμφόρησης, ε, να εστιάσουμε στα σημεία που πρέπει να ρυθμίζονται και να διέπονται από κανόνες κτλ. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να έχουμε και ασύμετρη νομοθεσία και κανόνες ασύμετρους κανόνες, αλλά κάποια βασικά πράγματα που έχουν ε, αποδείξει την αξία τους να τα κρατήσουμε. Ε, μια τελευταία παρατήρηση για το 5G, για το 5G. Πολλοί ευρωβουλευτές ε, εντόπισαν τα σωστά προβλήματα. Υπάρχουν πολλές αμφιβαιότητες δηλαδή για το 5G. Υπάρχουν πολύ πιθανοί φραγμή και ίσως έλλειψη κινήτρων από κάποιους ε, παρόχους, κάποιες κατηγορίες ε, παρόχων να το αναπτύσσουν γρήγορα. Η Ήτρε έχει ετοιμάσει και μόλις εξέδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση όπου μιλάει για το πρόβλημα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και ένα από τα συμπεράσματα που αναφέρει αυτή η έκθεση και με τα οποία συμφωνώ απόλυτα είναι ότι σε ορισμένε περιπτώσεις ίσως θα ήταν χρήσιμο να επιτρέψουμε και νέους φορείς να μπουν στην αγορά. Γιατί, μια και οι ήδη κατεστηγμένοι ε, πάροχοι ε, κινητής τηλεφωνίας, ας πούμε, ακόμα αποκομίζουν ωφέλη από το 4G ή μπορεί να μην ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο 5G λόγω των αβεβαιοτήτων, ε, να επενδύσουν γρήγορα, καλό είναι να επιτρέψουμε νέους, σε νέους, α, νέες εταιρείες να μπουν στην αγορά. Στου επόμενου μήνε θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα του κώδικα. Ε, συμμετρική νομοθεσία και κανόνες για την πρόσβαση στους πόρους, ε, βασικά στο φάσμα δηλαδή. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία που έχετε στα χέρια σας που μπορούν να δημιουργήσουν τα σωστά κίνητρα για νέες κατηγορίες ε, operator να μπουν στην αγορά. Οποιασδήποτε φύσης, έτσι, ή οποιος, οποιοδήποτε operator να μπουν στην αγορά και να σπρώξουν, να οδηγήσουν, να αναγκάσουν τους άλλους να επενδύσουν. Ευχαριστούμε κυρία Φελίξ Αντώνιο. Ο κύριος Φόξ. Thank you. try and cover off. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Καταρχάς, ε, οι χρήστες ε, δεν θέλουν την διακοπή, την διαταραχή ε, και δεν θέλουν υπερβολικές ρυθμίσεις γιατί αυτό αποτρέπει τις επενδύσεις και τους αποσπά από αυτό που πρέπει να κάνουν. Κατά τη γνώμη μας, τα περισσότερα, η ολοκλήρωση των δικτύων έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό, όμως υπάρχουν κάποια ζητήματα όσον αφορά την εξάπλωση των δικτύων. Ε, υπάρχει χώρος ε, και για τους μικρότερους φορείς και ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν πολύ μικρότεροι πάροχοι. Η αγορά είναι πολύ δυναμική και συνεπώς είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν ε, κατεστημένο φορέα εκμετάλλευσης, έναν κυρίαρχο φορέα, να κρατήσει μία ε, θέση ε, πρέπει να δούμε πού ακριβώς θα γίνει επένδυση, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και πολύ περιοριστικοί ως προς αυτό. Ε, με ρωτήσατε για το 5G και τον αντίκτυπό του. Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος ε, θα είναι ε, σταθμοί βάσης πολύ μεγάλη που θα είναι πάρα πολύ δαπανηροί και δεν είναι σαφές αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν αρκετά επιχειρηματικοί, ε, επιχειρηματικές περιπτώσεις που να μπορούν ακριβώς να ε, καλύψουν ε, αυτήν την, την, αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανένας άλλος που θέλει να κάνει ερωτήσεις στους προσκεκλημένους ομιλητές μας. Όχι. Ωραία. Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο τμήμα της ακρόασής μας, ε, με την ίδια σειρά, απλώς θα απαντήσουμε με την ε, αντίστροφη σειρά. Λοιπόν, να αρχίσουμε συνεπώς με τον κύριο Σοριάνο. Έχετε το λόγο. Το θέμα μας τώρα είναι αυτή τη φορά η διακυβέρνηση. Αυτό είναι το βασικό μας ε, ζήτημα τώρα. Κύριε Σοριάνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, όπως είπα και στο πρώτο πάνελ, εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε στην εφαρμογή των νέων στόχων που θα θέσουν ε, ε, τα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι πώς θα συμμετέχει ε, το ΜΠΕΡΕΚ ε, σε αυτήν την ε, σημαντική φιλοδοξία. Δύο ζητήματα. Πρώτον, ποιες είναι οι νέες αποστολές που θέλετε το ΜΠΕΡΕΚ να εκπληρώσει. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, χρειάζεται ένα νέο ΜΠΕΡΕΚ για να γίνει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τις νέες ε, αποστολές, ε, το Μπέρεκ ε, έχει αναφέρει ότι συμφωνεί, συμφωνεί με την ανεξαρτησία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και με τις, τα νέα καθήκοντα που θέλει να δώσει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές όσον αφορά το φάσμα, όσον αφορά τη χαρτογράφηση και τους τελικούς χρήστες εκτός από ε, την ασφάλεια των δικτύων, τον ανταγωνισμό κλπ. Νομίζω ότι συμφωνούμε ε, σε, βαθμό, σε μεγάλο βαθμό ως προς τις νέες αποστολές που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δοθούν στις νέες ε, ρυθμιστικές αρχές και το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει το Μπέρεκ. Το ερώτημα είναι τώρα αν χρειάζεται ένα νέο Μπέρεκ, ένα νέο φορέας ρυθμιστικών αρχών για να επιτυχθεί αυτό. Εμείς εκεί δεν, συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι το ΜΠΕΡΕΚ ε, είναι το αποτέλεσμα πολιτικών συζητήσεων ε, σε προηγούμενη αναθεώρηση και ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο δεν δραμάτισε σημαντικό ρόλο. Η κυρία Πιλάρ Δελκαστίγιο, ε, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και εκείνη. Ε, γιατί ο ρόλος του ΠΕΡΕΚ ε, είναι να συνεργάζονται οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές με ένα διοικητικό γραφείο που εδρεύει στη Ρήγα. Λοιπόν, Έχετε λοιπόν ε, ανθρώπους της δικής μου ομάδας, ε, ανθρώπους από την Ιταλία, από την Ουγγαρία που συνεργάζονται στην ομάδα πυρογνωμόνων για την αναθεώρηση. Το Μπέρεκ είναι ένας πολύ ιδιαίτερο συνδυασμός. είναι μια αποστολή ε, δέσμευσης. Εμείς είμαστε δεσμευμένοι στο να εξεύρουμε λύσεις από κοινού. Στο σύστημα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει ένας εκτελεστικός διευθυντής με τη δική του διοίκηση που θα είναι ουσιαστικά ένα, μια θηγατρική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα τα αποφασίζει όλα, θα τα προετοιμάζει όλα και εμείς ε, απλώς θα βάζουμε σφραγίδες στις αποφάσεις ως ρυθμιστικός φορέας. Δεν συμμετέχουμε όμως πλέον. Θα είναι μια νέα γραφειοκρατία. Δεν ε, θα... Δεν θα μας δοθεί το κίνητρο να κάνουμε κάτι μαζί, θα χάσουμε αυτήν την εθνική συμμετοχή. τι ξέρετε ότι στο ΜΠΕΡΕΚ όλες οι ομάδες ε, συγκεντρώνουν εθνικούς εμπειρογνώμονες που ξέρουν περί τίνος πρόκειται, γιατί εφαρμόζουν ε, τους κανονισμούς κάθε μέρα. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε ένα ιστορικό στο ΜΠΕΡΕΚ. Μου ζητήσατε, μας να επιβάλλουμε τον ανταγωνισμό, το κάναμε. Θελήσατε ε, ουδετερότητα των δικτύων και σχετικές προδιαγραφές τις είχατε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και η ε, κοινωνία των πολιτών τις επικρότησε. Δεν ήταν εύκολο ε, στην αρχή του εγχειρήματος αυτού. Επίσης, μερικές φορές διαφωνήσαμε μεταξύ μας ε, ως προς την εφαρμογή του πλαισίου Ξέρετε ότι έχουμε αυτή τη διαδικασία σε δύο φάσεις όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι ένας, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι δεν, ε, ένας ρυθμιστής δεν ε, πληρεί τις προποθέσει της. Ρωτά τον Μπέρεκ, συμφωνείτε. με το ότι εμείς διαφωνούμε με ε, την συμπεριφορά αυτού του εθνικού φορέα και κάθε φορά εμείς σχεδόν επιβεβαιώνουμε ε, την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία ομοτήμων, για να το πω έτσι, η οποία λειτουργεί και νομίζω ότι αν η προτεραιότητά σας είναι να χρησιμοποιήσετε το Μπέρεκ για να επιτύχετε τις, τους πολιτικούς σας ε, στόχους, ε, τότε ε, παρακαλώ μην τον καταργήσετε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να μεταρρυθμιστούμε, να μην καταπνίξουμε την ίδια μας τη δυναμική. Ευχαριστώ πολύ, πολύ ισχυρό μήνυμα. Κυρία Φύρ, Γενική Διευθύντρια, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για να σχολιάσω την διακυβέρνηση εγώ θα το κάνω από την πλευρά των χρηστών ε, και των τηλεπικοινωνιών. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι το καλύτερο, καλύτερος δείκτης και για τους χρήστες και για, τις, ε, ε, για τον τομέα. Βέβαια τα θεσμικά όργανα πρέπει να αποφασίσουν πώς θα γίνει αυτό. Παρόλα αυτά να μην σκοτώσουμε την κοινωνία Gigabit και ε, να, δώσουμε τη δυνατότητα ανάδειξης της ε, ε, καλύτερης συνδεσιμότητας σε ασύρματα δίκτυα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε εναρμόνιση του φάσματος, διαφορετικά δεν υπάρχει 5G και χωρίς το 5G δεν υπάρχει κοινωνία gigabit. Ε, το δεύτερο μου μήνυμα αφορά τη διαχείριση του φάσματος. Εμείς υποστηρίζουμε την εναρμόνιση της ε, διάρκειας των αδειών και πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητη συνιστόσα της ε, ύπαρξης κινήτρων ε, για επενδύσεις ε, στη μετάβαση στα νέα δίκτυα και πρέπει επίσης να τονίσω ότι ένα παραδοσιακό μοντέλο με μεμονωμένες άδειες πρέπει να αποτελέσει, να εξακολουθεί να αποτελεί το σκελετό του συστήματό μας. Και τρίτο και τελευταίο μήνυμά μου για τη διακυβέρνηση είναι ότι η ρυθμιστική απλοποίηση θα βοηθήσει το να υπερβούμε προβλήματα στον τομέα της διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι το σχέδιο μέτρων για την απλοποίηση της ανάλυσης της αγοράς πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και αυτό θα επέτρεπε όχι μόνο τις επενδύσεις αλλά και ανακούφιση ε, των πιέσεων για ε, ζητήματα διακυβέρνησης. Ε, όσο πιο απλή είναι και πιο προβλέψιμοι οι κανόνες, τόσο καλύτερη είναι η εφαρμογή και είναι και καλύτερη και ευκολότερη η δουλειά και των ρυθμιστικών, και των, ε, ρυθμιστικών φορέων και των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε εξασκηθεί, μου φαίνεται, ε, στο να δίνετε σύντομε ομιλίε. Είστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Κύριε Αντιπρόεδρε, Όλσον, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ εξίσου σύντομο με την προλαλή σα. Σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση τη ΠΕΡΕΚ, δεν νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο εμεί έχουμε να διατυπώσουμε άποψη. Αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουν οι εμπλεκόμενοι φορεί και θεσμικά όργανα. Ωστόσο, αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό ε, όταν συζητάμε για κανονισμούς και διακυβέρνηση και πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα, δώστε μου το μηχάνημα παρακαλώ. Αυτό που θα ήθελα εγώ να προκύψει από αυτή τη συζήτηση και όταν φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα για τη διακυβέρνηση. Αυτό που εγώ θέλω να δω είναι μια σχέση μεταξύ νομοθέτη και ρυθμιστή που δημιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο ε, θα οδηγήσει σε μια υποστηρικτική ε, νομοθεσία και, προ, και προνοητική. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, θα πρέπει να τα δούμε. Για παράδειγμα, δείτε σήμερα τι συζητούμε. Τις της εξελίξεις στο διαδίκτυο, στη τεχνολογία. Τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά για την κοινωνία συνολικά. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να προσαρμοστούμε πιο καλά στις αλλαγές που επισυμβαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί αυτή η ισορροπία μεταξύ νομοθέτη και ρυθμιστή, που θα επιτρέπει τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα. Και άλλα πράγματα, ε, τα προανέφερα όμως και δεν θέλω να τα επαναλάβω. Πάντω δράτω με τι ευκαιρίε, επειδή είμαι τόσο σύντομο σε αυτή τη δεύτερη ορολογία μου, να σχολιάσω ένα σημείο που νομίζω ότι είναι σημαντικό να τα ακούσει και η Επιτροπή σα. Η μελέτη που αναφέρθηκε πριν, την οποία είχατε αναθέσει ω Ήτρε, δεν συμφωνώ ότι είναι καλή για το 5G. Και το αντίθετο μάλιστα θα υποστήριζα ότι δηλαδή είναι μια μελέτη ε, που προσπαθεί να καλύψει τα πάντα, πάντο επιστητό, ε, δεν ε, πιστεύω ότι ο συντάκτης της μελέτης προβάλλει σωστά ε, το πόσο σημαντικό είναι να πετύχει το 5G στην Ευρώπη και μάλιστα υποβαθμίζει και το ρόλο της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Βιομηχανία. Σας δώσω έτσι ένα ε, στοιχείο. Ξέρουμε τι επενδύσεις κάνουν ε, οι φορείς εκμετάλλευσης. Αν δούμε τι θα γίνει το 2022. 25% κατά την ε, εκτίμησή μας ε, του τον είπα θα έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές 5G, 10% θα είναι το αντίστοιχο ποσό στην Ευρώπη, άρα κάτι πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Κύριε Φέλιτσο Αντώνιο. Από το Fast Web. Πιστεύω ότι το ισχύον σύστημα διακυβέρνησης μεταξύ της ΜΠΕΡΕΚ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, αποδείχθηκε πολύ ισορροπημένο και αποτελεσματικό στο παρελθόν. Η ανεξάρτησία των ε, ρυθμιστικών αρχών είναι πάρα πολύ σημαντική. Προφανώς είναι πιο σημαντική για τους μικρούς παρόχους ε, στο ίντερνετ παρά για τους μεγάλους. Προφανώς. Εμείς θέλουμε να είναι ισχυρές οι ρυθμιστικές αρχές για να μπορούν ανεξάρτητα να αξιολογούν τις συνθήκες της αγοράς και να ρυθμίζουν. με βάση τα τεχνικά στοιχεία. Είμαστε απόλυτα υπέρ της πρότασης της Κομισιόν να ενισχύσει τα κριτήρια ανεξαρτησίας και το προφίλ των ε, διευθυντών, των επικεφαλής δηλαδή των ρυθμιστικών αρχών. Είναι κάτι επιθυμητό. Εν συνεχεία, είμαστε υπέρ της εναρμόνισης και όχι της τυποποίησης. οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διατηρήσουν το δυναμικό και τις εξουσίες τους, να προβλέπουν τα κατάλληλα ένδικα μέσα και τις κατάλληλες υποχρεώσεις ε, με βάση την εθνική πραγματικότητα. Αυτό ήταν σημαντικό στο παρελθόν για να δοθεί όθηση στον ανταγωνισμό, για να προστατευτούν οι χρήστες και να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για καινοτομία. Τα κράτη-μέλη διαφέρουν πολύ το ένα από το άλλο. Και αυτό που στο ένα κράτος μέλος λειτουργεί, δεν λειτουργεί κατά ανάγκη σε όλα. Αυτή η φάση που διανύουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Η μετάβαση προς την κοινωνία των gigabit είναι πάρα πολύ σημαντική και δημιουργεί μεγαλύτερες διαφορές ε, στις προϋπάρχουσες καταστάσεις. Θέλουμε μια ισχυρή BEREC, με έναν ισχυρό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό φορέα, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρότερη ψηφιακή ενιαία αγορά στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φόξ, Ράμλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, η δομή της ε, διακυβέρνησης των ρυθμιστικών αρχών είναι πάρα πολύ περιπλοκό θέμα. Οι ε, επενδυτές ε, εστιάζουν στο αποτέλεσμα τη ρυθμιστικής διαδικασία και δηλαδή κρίνουμε βάση το αν ε, προωθούν τι επενδύσει, αυτά τα ρυθμιστικά πλαίσια ή όχι. Υπάρχουν τρει τομεί ε, που θα ήθελα να σχολιάσω. Καταρχάς, ε, κάτι θα σα είναι οικείο. όποιο και είναι το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι επενδύσει. Αυτό θα πρέπει να αναγνωστεί ω βασικό στόχο. Δεύτερον, ε, κάποιες από τι προκλήσει για την για το να, να μπορούν οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές να λάβουν υπόψη την ε, εθνική πραγματικότητα και ε, καταμερισμός του φάσματος. Επίσης, ε, οι πανευρωπαϊκοί φορείς όπως ο Μπέρε και η Κομισιόν θα πρέπει ε, να υιοθετήσουν ως στόχο ε, την δημιουργία ε, αποτελεσματικών επενδύσεων στο δίκτυο. Ε, αν αναπτυχθούν αποτελεσματικά ε, και συντηρηθούν και αναβαθμιστούν οι υποδομές των τηλεπικοινωνιών, αυτό θα είναι σωστό ε, είναι καλός, θα πρέπει να είναι σαφής στόχος της εθνιστικής πολιτικής ε, και με αυτόν τον τρόπο ε, θα μειωθεί και το μοναδιαίο κόστος των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Δεύτερον, είναι δύσκολο να δώσουμε μια οριστική απάντηση. Οι επενδυτές είναι ευαίσθητοι στην ιδέα ότι αλλάζουν οι συνθήκες από αγορά σε αγορά, ενώ τα οικονομικά στοιχεία είναι δεδομένα ε, όποια και είναι το κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να προωθήσει τις επενδύσεις. Ε, θα πρέπει να γίνουν κάποιες συστάσεις ε, χωρίς διακρίσεις. Ε, σε ορισμένε ε, περιπτώσεις οι τιμές των οπτικών ινών ε, συνδέονται, γίνονται, καθορίζονται μετά από έλεγχο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ε, δεν έχουμε σταθερότητα. Ε, το, βασικό είναι να έχουμε ε, καλύτερα αποτελέσματα, ε, υψηλότερη ταχύτητα και βελτιωμένη ε, ποιότητα στις υπηρεσίες. Ε, θα πρέπει να υπάρχει και συνέπεια και ποικιλομορφία. Η συνέπεια ε, δίνει δυνατότητα στους ε, παρόχους να αξιολογήσουν τις δυνατότητες που έχουν σε διαφορετικές αγορές, ε, μπορούν να κάνουν τοπικό πειραματισμό, μπορούν να υπάρχει ανταγωνισμός στις διάφορες κανονιστικές προσεγγίσεις και μπορούν να επιλέξουν την καλύτερη λύση. θα πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός προσαρμοστικότητας στις τοπικές συνθήκες, αλλά το πρόβλημα είναι όταν υπάρχει ουσιαστική απόκληση από τις βασικές αρχές ε, όταν υπάρχει όμως μεγαλύτερη ποικιλομορφία, όχι στις αρχές της ε, ρύθμισης, αλλά στην εφαρμογή της, ε, θα πρέπει να υπάρχει μόνο και μόνο για να απεικονίζονται οι περιφερειακές διαφορές στις αγορές. Ε, είναι σημαντικό οι τοπικές ε, ρυθμιστικές αρχές να λάβουν υπόψη τους τον υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας στις αστικές περιοχές. Το φάσμα τελικά. Τρεις είναι οι επιθυμίες των επενδυτών. Καταρχάς, θα πρέπει να δοθεί αρκετό φάσμα ε, οι οδικοί χάρτες ε, βοηθούν τους ε, operator των δικτών να σχεδιάσουν τις πολύ σημαντικές επενδύσεις και τα ποσά τα μεγάλα που πρέπει να πληρώσουν. όταν ένας operator δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, ε, υπάρχουν πολλοί πολλαπλοί διαγωνισμοί. Είναι σημαντικό να υπάρχει ε, συντονισμός και σαφήνεια. Ε, επίσης θα πρέπει να γίνουν δημοπρασίες του φάσματος με διαφανή και συνεπή τρόπο, ε, ούτως ώστε να υπάρχει προβλεψιμότητα. Ε, το φάσμα και οι επενδύσεις στις υποδομές ε, συνδέονται μεταξύ τους. Ε, εάν πληρωθεί ψηλή, την, ψηλή τιμή για το φάσμα, θα υπάρχει λιγότερο κεφάλαιο διαθέσιμο για να βελτιωθεί το δίκτυο. Τέλος, ε, το επεκτείνουμε τη διάρκεια των αδειών αυτό δίνει μεγαλύτερη βεβαιότητα μακροπρόθεσμα, ενώ ε, μπορούμε ε, να χορηγούμε το σπέκτρου με όρους αγοράς. Δηλαδή να λάβουμε υπόψη μας ότι το φάσμα είναι ε, ένα εμπορικό αγαθό. Επίσης θα πρέπει ό,τι και να κάνουμε σε κανονιστικό επίπεδο να αναγνώσουμε τη, τη σημασία της όθηση που πρέπει να δοθούν σε επενδύσει. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ισορροπία ανάμεσα στου τοπικού φορεί και στην, στο κανονιστικό πλαίσιο. Και αν ο, το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι προβλέψιμο, τότε θα μπορέσουν να κάνουν τι τεράστιε επενδύσει που χρειάζονται οι επενδυτέ. Ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα που δεν το συζητήσαμε και συγκεκριμένα η δορυφορική ευρυζωνικότητα. Έχουμε εκπροσώπους, από όσων γνωρίζω, από την Ένωση, ε, την κυρία Άρτιο Χόλα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δορυφορικών και από τη Utelsat έχουμε εκπρόσωπο. Δεν ξέρω αν ε, οι δύο θέλουν κάτι να πούν. Πολύ σύντομα όμως, ε, γιατί σε ό,τι αφορά την δορυφορική ευρυζωνικότητα, και την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ε, είναι καλό να ακούσουμε την άποψή σας πριν ε, ερωτήσουν οι βουλευτές. Κυρία Αρτιχόλα, European Satellite Operators Association, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε ότι οι επενδύσεις είναι το βασικό εδώ και πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που ε, θα προσελκύσει στα μελλοντικά δίκτυα ιδιωτικέ επενδύσεις. Ε, οι πραγματικοί περιορισμοί που υπάρχουν σήμερα για τις επενδύσεις σημαίνει ότι μόνο η αστική ελίτ ε, επωφελείται και όταν είμαστε σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι πιο κοντά στους πολίτες της, και είναι και φωνή της ε, το Κοινοβούλιο ε, και περισσότερο θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η προσβασιμότητα. Θα έπρεπε λοιπόν ο κώδικας να μιλά για ένα μείγμα τεχνολογιών, να υπάρχει καθολική υπηρεσία. Η οπτική είναι σίγουρα είναι η ιδανική λύση, αλλά αν ο κώδικας εστιάζει μόνο ε, στις οπτικές ίνες για το 5G, τότε το ψυχιακό χάσμα, το 5G θα γίνει χάος, θα γίνει άβυσος και Επίσης θα πρέπει να προωθηθεί εδώ ένα μείγμα τεχνολογιών αλλά με βάση την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. Έρχομαι τώρα στην δορυφορική ευρυζωνικότητα. Τα voucher schemes θα πρέπει να περιληφθούν στην αναθεώρηση των σχεδίων ευρυζωνικότητας. Είναι κάτι το οποίο ενθαρρύνει ε, την ευρυζωνικότητα στην Ήπεθρο. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι σήμερα βασίζονται ε, στην τηλεόραση, στην ε, χρήση δεδομένων, είτε άμεσα είτε έμεσα. Αυτό παρήχεται από δορυφόρου και 100% επενδύσει εδώ είναι ιδιωτικέ. Ε, στο αεροδρόμιο, στη θάλασσα, στα σπίτια, για λόγου ασφάλεια. Επομένω, διατάξει για το φάσμα θα πρέπει να αναφέρουν και την προστασία των κατεστημένων αυτών υπηρεσιών και όχι μόνο για να συνεχίσουν να παρέχουν οι πάροχοι αυτής τη υπηρεσία, αλλά και για ε, το ότι αν ε, δεν υπάρχουν αυτά δεν θα πληρώσουν οι χρήστε για βελτιώσει ε, τεχνολογία τεχνολογίας ή ξέρω εγώ για ενσωμάτωση συστήματο αυτοκινητών του, εφόσον αυτό δεν θα λειτουργεί παντού. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριο τώρα Στέφανο Αντωνέλη από τη Utilsat. Ευχαριστώ πολύ. Υπόθηκε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο ψηφιακό χάσμα στις περιοχές επεξεργασίας. Αυτό θα πρέπει να το ε, εκκριζώσουμε. Με τις προβλεπόμενες, εντάξει, νομίζω ότι δεν καλύπτονται τα πάντα. Θα πρέπει να λυθούν και άλλα μέτρα. Θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη βριζονικότητα, ιδίω στην Ήπεθρο και στι απόμακρε περιοχέ. Τρία στοιχεία. Το ένα αναφέρθηκε, τεχνολογική ουδετερότητα, θεμελιώδη αρχή. Εξίσου σημαντικό είναι όμω όχι μόνο να προωθηθεί ένα μείγμα τεχνολογιών, αλλά να βρεθούν και βρεδικέ λύσει που θα βασίζονται δηλαδή σε συνδυασμού διαφορετικών τεχνολογιών για την παροχή υπηρεσιών. Δεύτερον, υψηλή ποιότητα συνδεσιμότητα για την ύπεθρο για τι αγροτικέ περιοχέ. Ο στόχο είναι η σύνδεση επίση των δυνατών περισσότερων πόλεων στο λιγότερο χρονικό διάστημα ε, και με τις πιο προηγμένε τεχνολογίες. Ε, οι ποιοτικέ παράμετροι δεν είναι μόνο ε, η γρήγορη ταχύτητα μεταφόρτωση. Επίσης, καθολική υπηρεσία. Όχι μόνο για τις ευάλωτε ομάδε όλου όλους πολίτε που ε, υποφέρουν από το ψηφιακό χάσμα. Και οι προσιτές τιμές και η, διαθεσιμότητα λοιπόν είναι σημαντικά. Η δορυφορική τώρα βρυζανικότητα είναι μια ρεαλιστική λύση. Ήδη έχει επιτευχθεί ο στόχος το 2013. Και πάμε σε τον επόμενο στόχο, είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε προβλήματα στις επενδύσεις οι δορυφόροι λειτουργούν ίσως με διαφορετική αρχιτεκτονική από τις άλλες τηλεπικοινωνίες, όμως παρέχουν πολύ καλές υπηρεσίες. Πρόεδρος, ε, να έλθω στους εισηγητές μας. Η κυρία Ντελκαστίγιο, θέλετε το λόγο ή όχι. Για την Πέρεκ, θέλετε να ξεκινήσουμε από την Πέρεκ. Εντάξει, κύριο Σταχτουσενόφσκι, να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις παρουσιάσεις που ήταν σαφέστατες. Γιατί πιστεύω ότι η δική σας άποψη συμφωνεί με τις απόψεις πολλών συναδέλφων και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Μπέρεκ, πάντοτε αποτελούσε έναν διεύλο επικοινωνίας ε, ιδιαίτερα σημαντικό ανεξάρτητο και μπορώ να πω ότι σε πολλές περιπτώσεις, στην περίπτωση της ενέργειας για παράδειγμα, θα χρειαζόταν ε, έναν τέτοιου είδους οργανισμό. Θα του ήταν πολύ χρήσιμος. Και θα ήθελα να, ζητήσω από, να, να ρωτήσω όλους τους ε, προσκεκλημένους ποια είναι η άποψή τους για τον Μπέρεκ. Ίσως όμως έτσι Ίσως όμως θα μπορούσε να δοθεί αυτή η απάντηση και των θυρών. Θα ήθελα στη Γενική Διευθύντρια να θέσω το εξή ερώτημα. Αναφερθήκατε στις νέες αρμοδιότητες, τα νέα καθήκοντα όσον αφορά τις ε, βασικές αρμοδιότητες ε, οι οποίες κατά τη γνώμη σας, κατά το νέο αυτό στάδιο, αν υπάρξει ε, η έγκριση του κώδικα, και βάσει του τεχνολογικού προφίλ που αναδύεται μπροστά μας με τις νέες τεχνολογίες, θα μπορέσουμε να άρουμε τα εμπόδια που μπόρεσε να εντοπίσει τον ΠΕΡΕΚ στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν πώς, είναι, πώς διαφαίνεται ο ρόλος του ΠΕΡΕΚ στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής. Η κυρία Ντελκαστήλιο. Ευχαριστώ πολύ. Για αυτό το ζήτημα της διακυβέρνησης, ε, εντάξει, υπάρχουν δύο στοιχεία, οι υπηρεσίες από τη μία, η διαχείριση του φάσματος από την άλλη. Ε, Όσον αφορά το φάσμα, εγώ δεν θα πω πολλά. Γιατί πρέπει να πω ότι το Κοινοβούλιο συνάδει πλήρως με όλα αυτά που είπατε. Και άλλωστε φάνηκε και ε, στην ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών και το σχετικό κανονισμό. Ο κύριος Fox Romley αναφέρθηκε ε, διεξοδικότατα σε αυτό και ε, δεν συμφωνούμε, είμαστε στο, στο ίδιο μήκο το ερώτημά μου όμως είναι το εξή. Κύριε Σοριάνο, επικεφαλής του Μπέρεκ, αναφερθήκατε στο ότι χρειάζεστε μια νέα πνοή. Νομίζω ότι το Μπέρεκ ε, με εξαιρετικό τρόπο έχει εκπληρώσει την ε, αποστολή του και ανταποκρίθηκε στην έκκληση ε, στις εκκλήσεις που του έγιναν όταν ξεκίνησε το έργο του. Όμως, Ίσως θα μπορούσαμε να ήταν ενδιαφέρον αυτό, να υπάρξει ένας, ε, μία σύνδεση με τις τοπικές ε, αγορές ε, για την επίτευξη των κοινών στόχων και τον εντοπισμό των κοινών αναγκών. Αυτό είναι μία νέα πνοή. Αυτό το double lock που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε όταν εθνικός ρυθμιστής ε, δεν παίζει το ρόλο που πρέπει για να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να αποτελεί ένα εμπόδιο για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Αυτό όμως δεν είναι μια περίπτωση που καλύπτεται, από αυτήν τη μεταρρύθμιση στην οποία αναφέρεται και τη νέα πνοή που χρειάζεστε. Εννοώ τις τοπικές αγορές και το γεγονός ότι πρέπει να καταστεί πραγματικότητα η ψηφιακή ενιαία αγορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζουρίνιο, εισηγητής για το Wi-Fi for Europe. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες τελικά φαίνεται να είναι πολύ δυσκίνητες και γραφειοκρατικές ε, για την εφαρμογή, για τις διαδικασίες υλοποίησης. Η εν λόγω πρωτοβουλία Wi-Fi for Europe ε, είναι και ένα πιλωτικό σχέδιο, που θα έπρεπε να είναι και πιλωτικό σχέδιο και ως προς την διακυβέρνηση. Πρέπει να είναι αξιόπιστο συμπαγέ σύστημα και όλη η διαδικασία θα πρέπει να βασίζεται στην αυτορύθμιση, αλλά και στην εμπιστοσύνη. Διότι εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε 6 με 8.000 συνδέσεις σε όλες τις χώρες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με 20.000 ευρώ τιμή ε, κατά κεφαλήν και έχουμε και όμως και τα διαφορετικά ταμεία που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Αν όμω θέλουμε να είμαστε και στην αιχμή τη τεχνολογίας, αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα θα πρέπει να αποδείξει ότι από τεχνολογικής πλευράς λειτουργεί, αλλά και από διοικητική πλευράς ότι είναι εφικτό να υλοποιηθεί. Άρα θα πρέπει να είναι υψηλό επίπεδο και να το εμπιστευτεί ο κόσμος που θα ε, μας επιτρέψει έτσι να ανοίξουμε νέους δρόμους και να αντιμετωπίσουμε και τη γραφειοκρατία. Θα ήθελα να ακούσω όλους τους ε, ομιλητές μας. Ποια είναι η άποψή τους. Μπορούμε να έχουμε ένα μοντέλο αυτορύθμισης και πώς θα είναι αυτό αξιόπιστο. Κύριο κύριος Μπόνι που είναι υπεύθυνο για το 5G. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σοριάνο γιατί έδωσε ένα σαφές μήνυμα για τη συζήτηση αυτή η εναρμόνιση των αποφάσεων που σχετίζονται με το φάσμα είναι σημαντική για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G. Και φυσικά μπορούμε να μιλούμε για κάποιες ε, συγκρούσεις, ε, αντιπαραθέσεις, αλλά πρέπει να μπορούμε να κατανοούμε και τις απόψεις μας εδώ. Το μοντέλο που, υπάρχουν, που υπάρχει στη BEREC και στους θεσμούς της BEREC είναι bottom-up. Οι τεχνικοί επεξεργάζονται λύσεις. Η πλέον καστίγιο ανέφερε μια δυνατότητα, που θα μπορούσε να είναι και η συμβιβαστική λύση. Πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε το καλύτερο δυνατό μοντέλο εναρμόνισης για την κατανομή φάσματος. και δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι δεν υπάρχει μόνο η ΡΕΕ, η Μπέρεκ, οι φορείς εκμετάλλευσης και τα λοιπά στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν και τα κράτη-μέλη και Πολλές χώρες θα ε, θέσουν ε, καυτά ερωτήματα. Άρα το επόμενο βήμα για τη σημερινή συζήτηση είναι πώς θα υπάρξει αυτή η διακυβέρνηση των διαδικασιών με τη συμμετοχή των κρατών μελών. Πώς θα τα πιέσουμε, το λέω ανοιχτά τα κράτη-μέλη. Πώς θα τα πείσουμε ότι είναι σημαντικό. Ότι πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις ταυτόχρονα, γιατί για την υλοποίηση του 5G αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ τώρα κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Μία ερώτηση έχω μόνο. Και ε, για να είμαι βέβαια ότι κατάλαβα πολύ καλά με βάση αυτά που είπατε. Νομίζω ότι συμπεραίνω τη στόλη υπέρ της αναρμόνησης. Και αν δούμε και την εργαλειοθήκη, θα πρέπει να υπάρξει συντονισμό. Δεν άκουσα να λέει κανεί όμω ότι χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό οργανισμό. Κατάλαβα καλά. Δεν άκουσα κάποιο που να ε, υποστηρίζει τη δημιουργία ενό ευρωπαϊκού οργανισμού. Εκτό αν δεν το κατάλαβα ή μου ξέφυγε. Αλλά θα ήθελα μια σαφή απάντηση. Με Τα κράτη-μέλη ε, επί ε, τα συζητούμε όλα αυτά και πρέπει να δούμε τι θα γίνει, να εναρμόνιση, πώ θα προχωρήσουμε, ποια είναι η εργαλειοθήκη κτλ. κτλ, κτλ. Υπάρχει όμως ε, επιμονή για τη δημιουργία ενός ε, ευρωπαϊκού οργανισμού. Εσείς ποια ε, άποψη έχετε από αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Κούμπουλα να... Πολύ σύντομη. Και θα πρέπει να φύγω γιατί έχω μία άλλη συνάντηση. Ε, δύο ερωτήματα μπορώ να μου απαντήσει στον Μπέρεκ. Αν δεν είναι πάρα πολύ δομημένο, πώς εξασφαλίζεται ότι εισακούονται όλοι οι τοπικοί ρυθμιστικοί φορείς, οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς. Γιατί παρουσιάζεται εσεί το σύνολο του Μπέρεκ, αλλά μήπως ε, ξέρω εγώ, έχουμε το Λουξεμβούργο από τη μία και τη Γερμανία από την άλλη. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο, από με μεγέθους είναι τελείως διαφορετικές αυτές οι χώρες. Θέλω να μου εξηγήσετε δηλαδή διασυνοριακά πώς λειτουργεί αυτό. υπάρχει ένα ρυθμιστικό φορέας, ε, ακόμη και αν είναι ένα διασυνοριακό θέμα. Πώς λειτουργεί αυτό. Επίσης δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά ε, σε σχέση με το τι Ακριβώ είναι ο ρόλος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά πόσο μπορεί να τον εκχωρήσει αυτόν στον Μπέρεκ. Και μία άποψη, αν θέλετε, την ακούτε. Νομίζω ότι η εναρμόνιση ενέχει τον κίνδυνο να επιβραδύνουμε ε, την δυνατότητα των πρωτοστατών να κινηθούν πολύ γρήγορα γιατί θέλουν να κάνουν δοκιμές του 5G οι επιχειρήσεις. Ε, ήδη υπάρχει ένα νέο ε, φάσμα το οποίο έχει δοθεί Αν λέτε λοιπόν ότι όλοι ε, πρέπει να ε, κάνουν τη μετάβαση παράλληλα, ε, τότε δεν θα έχουμε ποτέ πρωτοστάτη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Κίνα πάει πολύ γρήγορα, άλλες χώρες πάνε πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορούμε να περιμένουμε πλήρη εναρμόνιση για να γίνει για να λειτουργήσει το σύστημα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω καμία άλλη ερώτηση. Αγαπητοί προσκεκλημένοι ομιλητές, μπορείτε να πείτε και μερικά πράγματα για τη δορυφορική ευρυζωνικότητα. Σε εσά επαφίεται. Κύριε Fox λέει, ε, από την Global Telecoms, αναλυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το θέμα των δορυφόρων. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι ε, η υποχρέωση οικομενικής ε, παροχής υπηρεσίας ε, για την ευρυζωνικότητα είναι πολύ σημαντική, όμως κάπως πρέπει να πληρώνεται και είναι δυσανάλογα ακριβή 5 με 10% εξάπλωση δικτύου στις ευρωπαϊκές χώρες, οπότε η αγορά πρέπει να υπαγορεύει ποια θα πρέπει να είναι η θέση και Πιστεύω ακράδαντα ότι το αποτέλεσμα θα, ήταν, θα είναι καλύτερη η ποιότητα. Ε, η, η, η, του δικτύου λοιπόν είναι πολύ σημαντική ως προς αυτό. Ε, όπως είπα, οι επενδυτές έχουν δεν έχουν πλήρεις ε, εμπεριστατωμένε ε, απόψεις ακόμη. Νομίζω ότι ε, το Μπέρεκ παίζει έναν χρήσιμο και σημαντικό ρόλο εκπροσωπώντας διαφορετικές καταστάσεις ρυθμιστικών φορέων στις Βρυξέλλες. Όμως πρέπει και οι εθνικοί ρυθμιστικές αρχές να μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις εμπειρίες τους ε, στον ΠΕΡΕΚ. Νομίζω λοιπόν ότι το επίπεδο της τοπικής εμπειρογνωμοσύνης είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό, αυτό είναι επιχείρημα κατά του ευρωπαϊκού ρυθμιστή ε, της ρύθμισης δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο. Ευχαριστώ πολύ μπορείτε να αναφερθείτε και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο θεωρείτε ότι δεν έχετε καλυφθεί για το, για το, για το πρώτο πάνελ. Εγώ... Θα ήθελα και εγώ σύντομα να κάνω και τα σχόλια, η κυρία Φελτσαντών, για κάποια ζητήματα τεχνολογικά και συμφωνώ με τον κύριο Φόξ Ράμλι 100% όταν λέει ότι υπήρξε κατά πάσα πιθανότητα, ιδίω σε κάποια κράτη-μέλη, ε, μεγάλο συνδεσιασμός με, τα, με τις οπτικές ε, ίνες και δόθηκε πολύ σημασία στο να φτάνουν αυτές μέχρι το σπίτι, μέχρι το νοικοκυριό. Και εγώ είμαι υπέρα, αλλά τέλος πάντων, fiber to the home δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι η λύση παντού, δεν μπορεί να είναι πανάκια, δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, θέλω να σας παραπέμψω για μια ακόμη φορά στην έκθεση που ανέθεσε η Επιτροπή Ήτρε για το 5G. Ένα σημαντικό πόρισμα της έκθεσης είναι ότι το ίδιο το 5G μπορεί να είναι εξαιρετικό υποκατάστατο ε, του fiber to the home για τις αγροτικές περιοχές και στη ΣΥΠΑ. Βλέπουμε ότι είναι άκρος ε, αποτελεσματικό και ξέρουμε ότι υπάρχει και υψηλό κόστος για την ομαλή ανάπτυξη του δικτύου στις αστικές περιοχές. Αυτό στο υπεθρό είναι διαφορετικό. Έρχομαι στο φάσμα, διαχείριση φάσματος, που συνδέεται στενά και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G. Νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό και το Κοινοβούλιο έκανε εξαιρετική δουλειά για τα φάσματα των 700 ε, τα κτλ. Θα πρέπει να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη ε, να ε, εφαρμόσουν τον λογικό οδικό χάρτη, το όραμα των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και η διαχείριση του φάσματος στον κώδικα εστιάζει επίσης και στους νεσερχόμενους φορείς και παρόχους. Διαχείριση φάσματος λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε να γίνει ένα σημαντικό μοχλός για την είσοδο νέων φορέων στην αγορά. Αυτό που χρειάζεται με το 5G η Ευρώπη είναι κάποιον επαναστάτη, κάποιον σκαπανέα ε, που έχει ε, ενδιαφέρον και πάρα πολύ γρήγορα θα αναπτύξει την τεχνολογία πιέζοντας έτσι και τους υπόλοιπους και το υπόλοιπο σύστημα. Ένας τολμηρός λοιπόν ε, που θα πρωτοστατήσει χρειάζεται. Και νομίζω ότι με τα σωστά κίνητρα θα πετύχουμε και με το 5G. Ευχαριστώ. Κυρία Φούρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς πιστεύουμε ότι η εναρμόνιση του φάσματος είναι σημαντική. Και μιλάμε για τη διάρκεια των αδειών επίσης, που είναι επίσης πολύ σημαντική. Ε, υπάρχει δυνατότητα καλύτερου συντονισμού, χωρίς να πιέζουμε προς τα έξω αυτούς που κάνουν πρώτη την κίνηση ε, σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να είναι αυτή η παρενέργεια της εναρμόνισης για το Μπέρεκ. Το έχω πει και στο παρελθόν. Είναι πολύ σημαντικό το Μπέρεκ. Το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό της προσπάθειας. Δεν θέλουμε να ε, επιβραδύνουμε την ε, έλευση της κοινωνίας του Gigabit. Ε, από την άλλη όμως, εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει μία λύση για όλους. Δεν ξεχνάμε τις διαφορές που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη γεωγραφικός, τοπολογικός και από κάθε άποψη. Ε, ναι, μεν στην εναρμόνιση, αλλά τις διαφορές που να συλλάβουμε υπόψη. Ο κύριος Σοριάνο. Ευχαριστώ. Να απαντήσω στο ερώτημα που ακούστηκε για τις βασικές αρμοδιότητες ε, που πρέπει να έχουν οι εθνικές αριθμιστικές αρχές. Εμείς συμφωνούμε με τις ε, αρμοδιότητες που αναφέρει ο νέος κώδικας. Αυτός που ζητάμε επιπλέον είναι να έχουμε ε, ευρύτερε αρμοδιότητες για συλλογή πληροφοριών σε επίπεδο υπηρεσιών. Γιατί αν θα πρέπει να αποφανθούμε για νέες υπηρεσίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο, αν θα πρέπει να θεωρηθούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή όχι, θα πρέπει να μπορούμε να συλλέγουμε ευρέω πληροφορίες και να θέτουμε ερωτήσεις στους ανθρώπους, ούτω ώστε σε ανθρώπους που τελικά δεν θα ε, θεωρηθούν, ας πούμε, operator. Ε, οι αρμοδιότητες και εξουσίες που προβλέπει η Κομισιόν είναι λίγο στενές προς το παρόν. η κυρία Καστίγιο Τελπιλά. Αν θέλετε συντονισμό υπάρχουν δύο στάδια. Καταρχά, το να δώσουμε αρμοδιότητα στι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ. Και αυτό ε, ε, μας καθιστά συνομιλητή όλων αυτών των εθνικών αρχών. Το να, του δίνουμε, να τους δίνουμε αρμοδιότητες, ε, αυτό είναι το ενακτήριο λάκτισμα για το συντονισμό. Αν μα δώσει δυνατότητα αύριο μεθαύριο να συμμετάσχουμε στην ε, κατανομή του φάσματο για τη διαμόρφωση τη αγορά, αυτό σημαίνει ότι αυτόματα ε, στον Μπερεκ θα συζητήσουμε αυτό το πράγμα και θα προσπαθήσουμε να επιφέρουμε μια κάποια εναρμόνιση. Θέλετε να πάτε πιο πέρα. Ε, και το θέμα του double lock, τι γίνεται με αυτό. Ε, δεν μου κάνει εντύπωση το ΜΠΕΡΕΚ, δεν θέλει κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε σύστημα double lock, ε, διπλού ε, δεν θέλουμε καθόλου περιορισμούς και εμπόδια. Σήμερα δεν μπορούμε παράλληλα να βάλουμε συστήματα πολύ περιοριστικά ε, στο επίπεδο της, του, κανονιστικού πλαισίου, ας πούμε, ε, και παράλληλα και να ασκήσουμε και βέτο, ας πούμε. Ε, τι περιθώριο ελιγμού θα έχουμε. Δεν θα πρέπει να είμαστε πολύ συντηρητικοί, θα πρέπει να τα δούμε τα πράγματα συνολικά και να δούμε αν οι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ έχουν την ε, αυτονομία για να βρουν λύσει σε εθνικό επίπεδο, ούτω ώστε να προωθήσουν τι επενδύσει, την ε, συνδεσιμότητα κλπ. Ευχαριστώ. Κύριε Όλσον. Αντιπρόεδρος της Έριξον. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάποια πράγματα που έχουν συζητηθεί ξανά εδώ. Το ρόλο των δορυφόρων, των δορυφορικών υπηρεσιών, το, οι δορυφορικέ υπηρεσίε είναι τμήμα του 5G. Έτσι θα είναι τμήμα του μελλοντικού ε, οικοσυστήματο οι δορυφορικέ εταιρείε. Υπάρχουν δυνατότητε ε, δορυφορικών ε, υβριδικών λύσεων, αλλά τελικά η αγορά θα αποφασίσει ποια είναι η οικονομικότερη και καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση. Επίση, το 5G τι ρόλο έχει ε, στη συνδεσιμότητα εναλλακτικά. Ε, αναφέρατε το τι συμβαίνει επίσης στις πολιτείες. Στις νομές ε, ε, βλέπουν, θα, συζη... χρησιμοποιήσουν το 5G για να συνδέσουν τα νοικοκυριά. Ε, από το κάμπινετ ως το σπίτι του χρήστη. Ε, στις υψηλότερες συχνότητες ε, καλό θα είναι να τις έχουμε στη διάθεσή μας για τη συνδεσιμότητα των οικοκυριών, για να έχουμε γρήγορο ίντερνετ. Τώρα, για τη συνδεσιμότητα και την ε, τεχνολογική ουδετερότητα. Οι, οι οπτικές ίνες ε, θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο για το 5G. Πολλοί δεν συνειδητοποιούν ότι η πλειοψηφία των base stations δεν συνδέονται με το καλώδιο, αλλά μέσω συνδέσεων point-to-point. -point. to point ότι σε κάνα ε, ε, δύο χρόνια, 2020, 2021, 2022, πάνω από τους μισούς base stations θα έχουν ε, microwave hops και θα έχουμε ταχύτητες πάνω από 10 gigabit. Ε, τέλος. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι θέλουμε να πετύχουμε και στο τι μπορούμε να πετύχουμε, αν θέλουμε να δώσουμε σε αυτούς που δεν είναι συνδεδεμένους την ε, εμπειρία της ε, κοινωνίας του Gigabit, δεν ξέρω θα συμβεί. Ε, ειδικά αν μιλάμε σε περιοχές που δεν έχουν σύνδεση αυτή τη στιγμή. Ε, για να του δώσουμε την δυνατότητα του Gigabit θα πρέπει να είναι καταρχά συνδεδεμένοι. Ε, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ε, base station και να περιμένουμε να του δώσουμε ταχύτητα του Gigabit ε, κατευθείαν. Ε, το θέμα είναι τι μπορούμε να πετύχουμε ε, και πώς και μπορούμε να το πετύχουμε με μια πλειάδα τεχνολογικών, τεχνολογιών μέχρι και του δορυφόρου. Οι δορυφόροι μπορούν να, δώσουν, να εξασφαλίσουν κάτι τέτοιο στι απομακρυσμένε περιοχέ πολύ πιο γρήγορα από ότι το Wi-Fi. Προσοχή, προσοχή λοιπόν. Το θέμα είναι πώς ορίζουμε τις λύσεις, τις τεχνολογικές λύσεις δηλαδή. Εναρμόνιση, δύο τελευταία λόγια. Είναι πολύ σημαντικό. Όπω είπε και η κυρία Κάμπελ, δεν μπορούμε φυσικά να επιτρέψουμε στους καθυστερημένους να παρεμποδίσουν την πρόοδο των πρωταθλητών. Αν μπορούμε με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν στην αγορά να μην σταματήσουμε περιοχές ή χώρες που θέλουν να κινηθούν πιο γρήγορα. Θα πρέπει να εστιάσουμε ε, στο να συμπεριλάβουμε τους πάντες, να μην υπάρξουν αποκλεισμοί, αλλά μην αφήσουμε και πολλούς και να καθυστερήσουν και να μας καθυστερήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική, ακριβή ε, ομιλία σα, επαγγελματικέ τα πάντα τα μάθαμε και τα ακούσαμε. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και μια σύντομη σύνοψη των, ε, από τους ηγητές. Στους οποίους απευθύνονταν στους τέσσερις αυτούς εισηγητές ε, οι παρεμβάσεις σας. Μισό λεπτό για τον κάθε εισηγητή, αν θέλετε να πει ο καθένας σας μία πρόταση. Είναι έτοιμος να πει κανείς το οτιδήποτε. Thank you. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Ντελκαστήγιο. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Ναι, κατάλαβα, δεν σα φτάνω τα 30 δευτερόλεπτα. Ωραία. Σα ευχαριστώ όλε και όλου. Ήταν εξαιρετική συνάντηση, εξαιρετική η ακρόαση. Θερμό ευχαριστώ σε όλου ε, του ομιλητέ μα. Συγχαρητήρια. Είστε επαγγελματίε, φαίνεται αυτό. Ευχαριστώ επίση του εισηγητέ. Ήταν πάρα πολύ καλή και οικοδομητική συνάντηση και για μένα που καθόμουν εδώ μαζί στο βήμα.